Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν συμφωνείτε, ξεκινήσουμε. Πρώτος ε, προσκεκλισμένος μας είναι ο Κάρλο Ριτσούτο, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ των Ερευνητικών Υποδομών, θα μας παρουσιάσει την έκθεση του 2009, που θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Έχουμε μέχρι τις 4 η ώρα για αυτό το θέμα και μετά συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Κύριε Ριτσούτο, έχετε τον λόγο. Ε, I ε, Θα προσπαθήσω να σας δώσω, ε, να σας ενημερώσω σχετικά ε, με τα τεκτενόμενα αυτού του φόρουμ. Ένας λόγος που έρχομαι ενώπιον της Επιτροπής εδώ του Κοινοβουλίου είναι διότι το Κοινοβούλιο μας στήριξε ιδιαιτέρως ε, στο παρελθόν. Στήριξε δηλαδή τις ε, προσπάθειές μας να εντάξουμε στην Ευρώπη αυτές τις υποδομές. Και μάλιστα ο πρόεδρος Μπούζεκ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών μας και διαρκώς μας πιέζει για δράση, για περαιτέρω δράση, κυρίως όσον αφορά ε, την εξισορρόπηση μεταξύ Ανατολής και Δύσης ε, στην Ευρώπη. Θα κάνω πρώτα απ' όλα μια σύντομη παρουσίαση του Φόρουμ. Δημιουργήθηκε το 2002 από το Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και ε, συγκεντρώνει εκπροσώπους από τα Υπουργεία ε, Έρευνας καθώς των κρατών μελών και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει την λήψη αποφάσεων και την στρατηγική προς την κινητοποίηση των τεχνολογιών, της έρευνας και την ενοποίηση της υποδομής έρευνας στην Ευρώπη. Ε, κοιτάξτε, έστω και αν ε, κάποια στιγμή δεν συμφωνείτε απολύτες ε, με όλα αυτά, το πιο σημαντικό που ε, κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τον τρόπο αυτό βλέπουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και επίσης φέρνουμε κοντά όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωση των κρατών μελών, των περιφερειών κτλ. Τώρα, ποιες είναι οι υποδομές έρευνας, γιατί μιλάμε δηλαδή. Πρέπει να πούμε ότι όλοι οι τομείς έρευνας χρειάζονται ε, προωθημένη ε, γνώση και βεβαίως υπάρχει ταυτόχρονα και η απέτηση τεχνολογικών, ε, τεχνικών απαντήσεων. Επομένως, εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε όλες αυτές τις επιστημονικές προκλήσεις ε, και τις τεχνικές απαντήσεις που σε αυτές θα πρέπει να δοθούν ε, είναι γεγονός ότι θα πρέπει όλες αυτές οι υποδομές να είναι ανοιχτές έτσι ώστε οι καλύτεροι, οι βέλτιστοι ερευνητές να μπορούν να συναντώνται η ολοένα μεγαλύτερη ικανότητα του τομέα πληροφορίας και επικοινωνίας απαιτεί πλέον και εξειδικευμένα εργαλεία. Εδώ σας δείχνω και μία διαφάνεια ε, για να σας δείξω ακριβώς με ποιο τρόπο βοηθάμε την επικοινωνία μεταξύ ε, των ε, επιστημονικών κοινοτήτων. Είτε πρόκειται για θέματα ενέργειας, είτε πρόκειται για θέματα γνώσης υλικών, είτε πρόκειται για κλιματολογικές συνθήκες. Οπωσδήποτε φέρνουμε κοντά τους επιστήμονες και τους βοηθούμε. Όταν ε, λειτουργούν λοιπόν ε, τα, ε, η δυναμική γνώση και τα τρίγωνα καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να, ελκύσουν, να ελκύουν την καινοτομία, την έρευνα καθώς επίσης και την καλύτερη γνώση και την τεχνολογία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε με σε αυτές τις ε, προκλήσεις ε, χρειάζομαστε να ε, φέρουμε κοντά όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό ελευθερώνουμε το δυναμικό το οποίο υπάρχει στον τομέα αυτό. Τώρα, εάν πρέπει να σας δώσω μία εικόνα αντί για ε, τρίγωνο έχουμε τη δομή του αδάμαντος. Ε, με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε να βελτιώσουμε την επαφή ανάμεσα στην, στους διάφορους παίκτες, είτε είναι τεχνολογικά Ινστιτούτα, είτε είναι πανεπιστήμια κτλ. Εάν λειτουργήσουν καλά όλα αυτά, φτάνουμε σε αυτήν την περίπλοκη εικόνα μέσω της οποίας αντί να έχουμε φυγή εγκεφάλων ε, μπορούμε να προωθήσουμε ε, τον, τον ε, επιστημονικό τουρισμό, την ανταλλαγή απόψεων και βέβαια μέσω και υψηλού επίπεδου δημοσίων διαγωνισμών. Είναι μια καλή οδός την οποία να ακολουθούμε. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η Γκρενόμπλ. Είναι το πεντάγωνο ή το πολύγωνο τέλο πάντων. Σε αυτήν την Χερσόνησο, νήσο, όπως να σας την πω. Τη δεκαετία του 70 λοιπόν αποφασίσαμε, αποφασίστηκε μάλλον ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί αυτή η στρογγυλή υποδομή που σας δείχνω τώρα, ε, το Ινστιτούτο Λόζεβέλ, που έχει από τότε ε, συμμετάσχει σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Πρόκειται για κάτι που δημιουργήθηκε από τρεις-τέσσερις χώρες μαζί. Μετά αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την άλλη υποδομή. Τώρα όλη αυτή η περιφέρεια, καθώς επίσης και περιοχές οι οποίες συνδέονται σε άλλα σημεία της Ευρώπης με αυτήν εδώ την περιοχή, ανθούν. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Πηγαίνοντας πίσω στο Μεσαίωνα, τα αβαία καθώς επίσης και κάποιες γνωστές ε, ε, βιβλιοθήκες But they Ανέπτυσαν ε, τεχνολογίες οι οποίες τότε ε, χρειάζονται έτσι ώστε να ε, μεταφερθεί η γνώση προς τα έξω. Και ανέπτυσαν μάλιστα και άλλες τεχνολογίες, χημεία, χημεία τρόφιμα, ποτά, αυτό το γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά τεχνολογίες οικοδομικές, κατασκευής, καθώς και άλλες τεχνολογίες τις οποίες ε, ε, ε, μετέδωσαν και προς την αναγέννηση. Επομένως, ξέρουμε ότι βοήθησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου και μάλιστα πολύ συχνά το επίκεντρο της αρχής ενός μιας εμπορικής διαδικασίας ήταν εκεί. Τώρα, κεντρικός πυλώνας στην ε, στην ΕΡΑ είναι ακριβώς η δήλωση ΛΑΝΤ του Ιουλίου 2009 ε, καθώς επίσης και η δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών του Φεβρουαρίου 2010. Ε, Πρόκειται για σημαντικές ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες ακριβώς δείχνουν όλα τα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία είναι παρόντα σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεμονωμένες χώρες δεν μπορούν να οικοδομήσουν ε, καθώς επίσης και να ε, ε, στηρίξουν την ανοιχτή πρόσβαση στα RI και επομένως ενώ έχουν μεγάλο δυναμικό πρέπει οπωσδήποτε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι υποδομές έρευνας να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ε, ε, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται και για ε, διαδικασίες οι οποίες απορροφούν πάρα πολλά χρήματα. Μπορεί να φτάσουν μέχρι 10-15 δις ευρώ. Μονάχα εάν ομαδοποιηθούν αυτού του είδους οι υποδομές έρευνας μπορούν ικανοποιητικά να χρησιμοποιήσουν τις νέες, τους νέους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως μπορούν να ανταποκριθούν ε, σωστά στις αναπτυσσόμενες προκλήσεις. Αυτές, η, ε, ε, αυτή η πρόκληση αναγνωρίστηκε σαφώς το 2000, το 2000 όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ΕΡΑ και το οποίο οδήγησε στη δημιουργία του ΕΣΦΡΙ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Όσον αφορά τώρα τις δραστηριότητες ΕΣΦΡΙ, εμείς ασχολούμαστε, ε, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τις ε, ε, περιφερειακές προοπτικές, κυρίως δε όσον αφορά την επανισορρόπηση Ανατολής και Δύσης. Επίσης ασχολούμεθα με την ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων, με την διαχείριση προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν όλους τους ενδιαφερόμενους κλπ. Η δράση μας ε, προετοιμάζεται από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια του δευτέρου προγράμματος ε, πλαισίου ε, και έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς και αναμειγνιόμεθα ιδιαιτέρως με ε, προγράμματα τα οποία ε, προωθούνται. Όπως ε, θα ξέρετε υπάρχει ένας νέος νομικός κανονισμός ο οποίος τίθεται σε ισχύ τώρα του Συμβουλίου και αφορά την νομική δομή που θα διέπει πλέον αυτές τις υποδομές. Ε, το θέμα επίσης στρατηγικής του 2020 είναι σημαντικό και εργαζόμαστε και γι' αυτό. Ε, τώρα, για τον οδικό χάρτη. Και πέρσι είχαμε παρουσιάσει ε, στην Επιτροπή σας τον οδικό χάρτη του ΕΣΦΡΙ. Εκεί έχουμε επιλέξει και καταδεικνύουμε 44 projects ε, ε, τα οποία επελέξαν μέσα από 200 προτάσεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ε, αυτός ο δικός χάρτης των 44 επιλεγμένων προγραμμάτων αποφασίστηκε ομόφωνα και επομένως και αυτό είναι ένα τμήμα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα αυξήσουμε, θα προσθεθούν κάποια ε, προγράμματα στον τομέα της, ε, της ε, υγείας, της ενέργειας και της διατροφής, των τροφίμων. 28 από τα 33 μέλη έχουν ήδη ανταποκριθεί μέσω εθνικών οδικών χαρτών, εκ των οποίων οι 13 έχουν ήδη δημοσιευθεί. Το σημαντικό είναι ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να οικοδομήσουμε κοινά ε, εργαλεία και για όλη την Ευρώπη. Βλέπετε εδώ ε, ότι ακόμα και νέες ε, χώρες μέλη έχουν εκπονήσει εθνικούς οδηγούς, οδικούς χάρτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Όσον αφορά την εφαρμογή τώρα του οδικού χάρτη, 10 νέα κέντρα ε, κέντρα έρευνας ε, εφαρμόζουν τώρα και, έχουν, και υπάρχουν πολλά άλλα τα οποία έχουν ήδη προχωρήσει πολύ περισσότερο. Άλλες εξελίξεις τώρα. Ε, εμείς καλύπτουμε σχεδόν τα πάντα. Όλες τις φυσικές επιστήμες, την χημεία, ε, ανθρωπιστικές επιστήμες ε, λοιπά Δημιουργούμε ε, επίσης εδεσμούς με κοινότητες οι οποίες δεν έχουν την κοινοτική σκέψη και δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με τον τρόπο αυτό. και βεβαίως ε, και περιφερειακά και περιφερειακοί διορθωτική πόροι χρησιμοποιούνται τώρα ε, για, την, ε, για τους Regional Partner Facilities έτσι ώστε, να ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως η... εμείς προσπαθούμε να... να μην έχουμε διαχωρισμό ανάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή, την κοινωνία ή την βιομηχανία βιομηχανία. Ε, ε, εμείς συνεργαζόμαστε επίσης ε, και με άλλες χώρες και με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία κτλ. Τώρα, είναι γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια, ε, έναν ευρωπαϊκό χώρο ε, έρευνας ε, μέσω των υποδομών έρευνας. Αλλά για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε και τις εθνικές και, τις, και τους εθνικούς και τους τοπικούς πόρους μέσα σε μια κοινή προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Και βέβαια βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη πιθανή πηγή ε, ε, επιπλέον χρηματοδότησης ε, για να καλυφθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αριστείας και, πρέπει, και, καλύπτει 20 με 30% των διεθνών προσπαθειών για το θέμα αυτό. Τα επόμενα βήματα τώρα είναι να έχουμε αηφορία, ε, βιωσιμότητα, ε, να δημιουργήσουμε ε, τον, τον ποιοτικό έλεγχο και βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους ανθρώπινους πόρους. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται ε, προσπάθεια ευρωπαϊκού επίπεδου έτσι ώστε να υπάρξει διαθεσμική ε, αριστεία ε, η οποία θα προσθεθεί στις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Έρευνας που αποσκοπούν στην ατομική ε, αριστεία και επομένως να δημιουργήσουμε μαζί με, την, με τις ε, τεχνολογίες μαζί ε, με το, και μαζί με τα JTIs έναν ευρωπαϊκό χώρο που θα αφορά όχι μονάχα την έρευνα αλλά και την καινοτομία. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για, τον, ε, για τη διαρκή σας προσπάθεια στήριξης και βεβαίως και για την άμεση στήριξη που μας παρέχετε και που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρεξ ζήτησε πρώτος τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ε, η μεγάλη πανευρωπαϊκή συγκέντρωση ερευνητικών δομών, οι, ε, διευρυμένε τέτοιε επαγγελματωμένε ε, ερευνητικέ δομέ μπορούν να προσελκύσουν ε, του νέου ερευνητέ και επιστήμονε και έτσι να παρεμποδίσουν τη διαρροή κεφάλων. Η δημιουργία τέτοιων ε, δομών θα πρέπει να συνοδεύονται από φύλλα πορεία που θα αναφέρουν αυτές τις υποδομές, γιατί οι υποδομές είναι πολύ δαπανηρές και η συντήρησή του το ίδιο. Επίσης, θα πρέπει να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επιστημόνων και των ερευνητών. Έτσι, όχι μόνο θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια αγορά, αλλά ε, θα ευνοηθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Βέβαια, θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσέγγιση αυτή κυβερνήση, ιδιαίτερα στις περιφέρειες της σύγκλησης. Πολλά αναφέρθηκαν από την έκθεσή σας για τα διαρθρωτικά ταμεία. Βέβαια, η κλίδα κατανομής των διαρθρωτικών ταμείων είναι διαφορετική. Πρόκειται για ένα νέο κανονισμό, ένα συμπληρωματικό κανονισμό. Γιατί στο, παράδειγμα, στο σημείο 4.3 των διαρθρωτικών ταμείων ε, προκύπτει από την έκθεση, ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά κονδύλια και τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα της ε, περίοδου 2007-2013. Αυτό αναφέρεται στο 4-3 της έκθεσής σας και αυτό με εκπλήσει γιατί αναφέρθηκε για την κατασκευή δρόμων υποδομής και οικολογικές ε, πρωτοβουλίες. Και είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοια δυνατότητα όπως αυτή που αναφέρεται στο 4.3. Θα ήθελα λοιπόν μια διευκρίνηση από αυτού. Και έχω μια ερώτηση. Υπήρξαν ήδη παραδείγματα αξιοποίησης ε, των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής προκειμένου να ενισχυθούν τέτοιες ερευνητικές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Μια και μιλούμε για υποδο, υποδομές είτε συγκεντρωμένες είτε εξαπλωμένες. Τι γίνεται με τα e-cities. Δηλαδή για τις ευφυείς πόλεις όπου το ερευνητικό πρόγραμμα και η ερευνητική υποδομή σε πειραματικό βέβαια στάδιο θα δοκιμαστεί ως ε, παγκόσμιο υπόδειγμα. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο υπόδειγμα. Γιατί ακόμη τέτοια ίση της δεν υπάρχουν στον κόσμο, οπότε με αυτήν την άποψη θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε πρωτοπόροι σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. κυρία Χέρτσογκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ριτσούτο. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ασχολείται με την έρευνα στην Ευρώπη αντιλαμβάνεται και σέβεται την εμπειρία σας και το πώς σκέφτεστε για την έρευνα για ολόκληρη την Ευρώπη. Παρά το ότι η Ουγγαρία δεν ήταν ε, μέλος της Ένωσης, ε, όταν αποφασίστηκε αυτή η οικονομία της γνώσης νομίζω ήταν κάτι καλό αυτό και νομίζω και το δίκτυο αυτό είναι συνέπεια της απόφασης αυτής. Ε, πρέπει λοιπόν να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρώτη μου ερώτηση όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 44 έργα στον κατάλογο. Πότε θα ξεκινήσει όμως το πρώτο, νομίζετε εσείς. Πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί κάτι και και να έχουμε αποτελέσματα. Κάτι άλλο που σας είπα και πριν στη συζήτηση που είχαμε, όταν κοιτάμε τις πιθανές τοποθεσίες ε, για αυτά τα, τα κλάστερ, νομίζω οτιδήποτε βόρεια από τα Πυρηναία είναι μια χαρά μέρος. Και Νομίζω πως έτσι το βλέπουν ορισμένοι καμιά φορά και αν είναι να μιλάμε για ανταλλαγή και όχι διαρροή εγκεφάλων πρέπει να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά. Αλλιώς η αλληλεγγύη δεν υπάρχει και κάποιες χώρες δίνουν και δεν ε, ε λαμβάνουν τίποτα για την ε, επένδυση που κάνουν και θα χάσουν αισιοδοξία τους και την στήριξη. Και ρωτάω για, κάτι, για ένα πολύ απλό λόγο. Εγώ έχω παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή και το τι έγινε και με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία και με άλλα ιδρύματα. Και υπάρχει μια τεράστια διαφορά γιατί εμείς τα είχαμε δει αυτά στην Ουγγαρία. Το ένα χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη, από τις χώρες ενώ το άλλο χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία. από τις νέες χώρες ε, δηλαδή, σε αντίθεση με κάποια άλλα έργα. Αυτές είναι οι βασικές μου λοιπόν ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου απαντήσετε πώς θα υπάρξει η ευρωπαϊκή Ελληνική και η ανταλλαγή εγκεφάλων και όχι η διαρροή εγκεφάλων. Για να μην πηγαίνουν όλα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Ρεζούτο για την πολύ ε, παραστατική του παρουσίαση του ΕΣΦΡΙ. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω σε, στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για την καθιέρωση του ενιαίου χώρου της έρευνας, των μεγάλων έργων υποδομών του ΕΣΦΡΙ, την ίδρυση του EIT, την ίδρυση του ERC. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη αποκτά μια αίσθηση ενότητος στην ερευνητική της προσπάθεια με όλα όσα και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ανέφεραν. Έχω την εντύπωση, η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Ριζούτο θα είναι ε, πολύ συγκεκριμένη. Η κυρία συνάδελφος που πριν μίλησε αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη στην έρευνα καθώς επίσης και σε γεωγραφική η διαρθρωτική κατανομή των πόρων της Ένωσης για τη διεξαγωγή έρευνας. Προέρχομαι από μια χώρα που δεν τη συμφέρει καθόλου να μιλάει για αριστεία, αλλά είμαι επιστήμων και πρέπει να θέσω το ζήτημα της ευρωπαϊκής έρευνας στη βάση του. Η ευρωπαϊκή έρευνα για την ώρα δεν αποτελεί την πρωτοπορία παγκοσμίω όπως είχαν φανταστεί το 2000 με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Οι εκδόσεις της Σουηδικής Προεδρίας με τον τίτλο European Paradise δείχνουν πολύ καλά ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και η αρχή της αλληλεγγύης ε, δεν είναι οι κατάλληλες αρχές για την ανάπτυξη παγκόσμια ανταγωνιστικής έρευνας. Συνεπώς, η επικέντρωση στην αρχή της αριστείας όπου και αν αυτή βρίσκεται στην Ευρώπη σε συνδυασμό με την μόνη αλληλεγγύη που γνωρίζω δηλαδή την μετακίνηση, την ελευθερία των ιδεών και των ανθρώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια είναι τα εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Η ερώτησή μου είναι πολύ σαφής κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε την εμπειρία αλλά και την ανασχόληση. Εάν ήσασταν ένας αξιολογητής του παγκοσμίου επιστημονικού συστήματος, πώς θα αξιολογούσατε τις υπάρχουσες υποδομές της Ευρώπης σήμερα, τις δυνατότητές της να παραγάγει μεγάλη επιστήμη, καθώς επίσης θα ήθελα να σας κάνω και μια αναπάντηχη ερώτηση, κατά πόσον πιστεύετε στις κατατεθειμένες, στους κατατεθειμένους οδικούς χάρτες που έχουν ε, κατατεθεί από τα κράτη-μέλη. Γνωρίζω ότι ο δρόμος της Ευρώπης για την οικοδόμηση από τον πολυπολιτισμικό και πολυεπίπεδο επιστημονικό της χώρο ενός ενιαίου χαρακτήρα που θα οδηγήσει σε παγκόσμιας φήμης επιστημονικές επιδόσεις παρόμοιες με αυτές της χρυσή τριακονταετίας των αρχών του 20ου αιώνα περνάει μέσα από μεγάλες προσπάθειες και θα ήθελα πολύ να μου πείτε εάν εσείς πιστεύετε ότι με, τους ακολουθούμε, με τις ακολουθούμενες προσπάθειες μεταξύ των οποίων και το ΕΣΦΡΙ στο οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ο κατάλληλος δρόμος για την Ευρώπη και για τους στόχους της. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Ριτσούτο για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και να πω ότι εδώ πίσω είμαι και όλα αυτά τα σχέδια και δραστηριότητες καθώς και το μελλοντικό όραμα του ΕΣΠΡΙ είναι ευπρόσδεκτα. Αναφερθήκατε σε τρεις πυλώνες καινοτομία. Αλλά αυτό που λείπει από εδώ είναι ο ρόλος της ανώτερης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην όλη διαδικασία. Σας ερωτώ λοιπόν, Πώς βλέπετε εσείς από τη θέση σας τη συνεργασία μεταξύ των ε, ε, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων, γιατί ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας γίνεται στα πανεπιστήμια και οι διδακτορικοί φοιτητέ ε, και στις διδακτορικές σπουδέ δίνεται ιδιαίτερος ρόλος σε αυτή τη διαδικασία. Πώς λοιπόν το φόρουμ σας μπορεί να προωθήσει αυτή τη συνεργασία και να εμποτίσει τα πανεπιστήμια με αυτή την οτροπία και τη στρατηγική για συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Ριτσούτο για την παρουσίαση της έκθεσής του και να θέσω δύο ερωτήσεις σε δύο σημεία που δείξατε ακροθυγώς. Μπορείτε να αναπτύξετε λίγο περισσότερο. Καταρχήν, τι γίνεται με τη μέσο και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αυτών των ερευνητικών υποδομών, που είναι, όπως είπαμε, πολύ δαπανηρές. Θα εξασφαλιστεί αυτή η μέσο και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, θα υπάρξει βιωσιμότητα αυτής της χρηματοδότησης, γιατί πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες στη χρηματοδότηση αυτή. Το δεύτερο θέμα το αναφέρατε προς το τέλος. Ποια είναι η σχέση των ερευνητικών υποδομών και των GTIs και ιδιαίτερα του IT που είναι νέο, νέος θεσμός. Βέβαια ασχολείται με θέματα ενέργειας, κλιματικών αλλαγών, την κοινωνία της πληροφορίας, ε, τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας. Ήδη υπάρχει συνεργασία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ε, οι ερευνητικές υποδομές από το IT. Ευχαριστώ κυρία Τούια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτήν την ε, ενδιαφέρουσα ε, την ενδιαφέρουσα παρέμβαση, την οποία δυστυχώ δεν άκουσα ολόκληρη. λαμβάνοντα υπόψη την βαθιά γνώση σα όσον αφορά θέματα έρευνα σε εθνικό και ε, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, θα ήθελα να σα πω κάτι το οποίο, να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν αφορά την ίδια την έρευνα, αλλά τα εργαλεία. Πώ δηλαδή μπορούμε να κάνουμε λειτουργική ε, αυτή την έρευνα και αυτά τα προγράμματα έρευνας. Γιατί έχω την άποψη ότι συζητάμε πολύ έχοντας στο νου μας κάποιους ε, μηχανισμούς που αρχίζουν να εφαρμόζονται έτσι ώστε ε, να έχουμε όλα αυτά τα ε, JTI, τις πλατφόρμες έρευνας κτλ. Αλλά αυτές οι διαδικασίες όλες, αντί να επιταχύνουν τις διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν προς αυτά αποτελέσματα, στην ουσία αποτελούν τροχοπέδι. Και επομένω ε, εσεί που συμμετέχετε σαν ΕΣΦΡΙ, δημιουργηθήκατε έτσι ώστε, το είπε άλλωστε και ο προηγούμενος αρμόδιος επίτροπος, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ένα ομοιογενές νομικό πλαίσιο ε, για να ε, δημιουργηθεί το κονσόρσιου μέρη. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα διαδικαστικά, προβλήματα οικονομικά κλπ. Είναι γεγονός ότι η επιλογή είναι πρόσφατη. Αλλά εγώ σας ρωτώ, λειτουργεί αυτή η επιλογή, θα λειτουργήσει. Ε, αν αυτό το εργαλείο, αντί εργαλείο ε, προώθησης, ε, τελικά μπορεί να καταλήξει επιβραδυντικός παράγων. Απ' την άλλη πλευρά, μας λένε και από τον τομέα της έρευνας και από τη βιομηχανία ότι αυτά τα JTIs δεν προχωρούν καλά. Και μια άλλη ερώτηση που έθεσε και η κυρία Καρβάλιο. Ε, ποιε είναι οι σχέσει σα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία, γιατί μερικέ φορέ και όσον αφορά τη σχέση αυτή έχουμε την αίσθηση ότι δημιουργούμε υπερβολικά πολλά, ε, υπερβολικούς, υπερβολικά πολλούς φορείς που τελικά κατακαιρματίζουν τον τομέα. Επομένως, εγώ ε, ρωτώ, όχι τόσο για την έρευνα, όσο για τα εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν την έρευνα αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει αρκετές ερωτήσεις ε, κύριε Ριτσούτο. Θα θέλαμε νομίζω κάποιες ε, απαντήσεις ε, και βεβαίως αναμένουμε μετά και την συμμετοχή των λοιπόν συναδέλφων. Λοιπόν, έχει τον λόγο. Ε... Καταρχήν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω εδώ και τον δόκτωρα Αντρέι Γιουνέλ, Ακρομανίας που είναι μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΦΡΙ. Δεν φανταζόμουν ότι θα έχω τόσες πολλές ερωτήσεις που αφορούν ε, την ισορροπία Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης. Αλλά νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ στην κατάλληλη θέση για να μας βοηθήσει να αντισταθμίσουμε τις υπάρχουσες ανισορροπίες. Θα προσπαθήσω εγώ να δώσω κάποιες απαντήσεις και αν ο Γιουνέλ θέλει να συμπληρώσει, πολύ ευχαρίστω. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση υπήρχε κυρίως ε, στις μεγάλες παλιές χώρες μέλη της Ένωσης. Και κατά κάποιο τρόπο υπήρχε μικρότερη συγκέντρωση στη Γερμανία από ό,τι στη Γαλλία υπήρχε αρχικά συγκέντρωση στα πιο παλιά, από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, θα μπορούσαμε να πούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί ξεκινήσαμε το χτίσιμο της Ευρώπης στη δεκαετία του 50. Αν πάρετε το ΣΕΡΝ, το ΓΕΣΕΡΕΦ και αν πάρετε κάποια από τα μεγάλα αυτά διεθνή κέντρα, είτε στηρίχθηκαν σε διακυβερνητική συνεργασία, είτε δημιουργήθηκαν και ιδρύθηκαν πριν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σημείο ιστορικής αναδρομής. Άφησα μία διαφάνεια, είχα αφήσει μάλλον, αλλά προς το, στο μεταξύ έχει εξαφανιστεί. Εν πάση περιπτώσει, οι χώρες που σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο είναι η Αυστρία, η Τσεχία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, Υπάρχει βέβαια και εκεί χάσμα. Η Λιθουανία, η Πολωνία. Και μάλιστα έμαθα ότι σήμερα το πρωί η Τσεχία αποφάσισε για 7 υποδομές. Υπάρχει λοιπόν κίνηση και πρόοδος. Δεν ήμουν ακόμη πρόεδρος του ΕΣΦΡΙ, αλλά με το που έγινε η διεύρυνση και εκεί υπήρξε κάποια αντίσταση, εγώ επιδίωξα τη διεύρυνση του ΕΣΦΡΙ πριν λάβει χώρα η διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς. Έγινε διεύρυνση ήδη σήμερα με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάτι άλλο που αφορά τη λειτουργία. Και τα οικονομικά ωφέλη. Το θέμα αυτό σχετίζεται με τις ερωτήσεις του κ. Τσουκαλά και της κυρίας Χέρτσοκ. Γιατί πολλά θέματα αναφέρθηκαν στο καταμερισμό, στην κατανομή όταν αρχίσαμε με το ΕΣΦΡΙ, η αρχική μας ιδέα ήταν να μιμηθούμε τις Ηνωμένε Πολιτείε καταρτίζοντας έναν οδικό χάρτη των ευρύτερων και πιο δαπανηρών ερευνητικών υποδομών. Αυτό που προωθούμε τώρα ως προσέγγιση είναι ότι δεν ενδιαφέρει το μέγεθος, δεν ενδιαφέρουν οι διαστάσεις, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει η ποιότητα. Η ποιότητα θα πρέπει να είναι απαράμιλη. Μπορεί να κοστίσει 10 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου. Και αν θέλουμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό, αυτό που συμβαίνει με τέτοιε ερευνητικέ υποδομέ είναι ότι είναι οι Ολυμπιακοί αγώνε τη έρευνα. Όταν, όταν διοργανώνουμε Ολυμπιακού αγώνε, η ποιότητα είναι Ολυμπιακή ποιότητα, άσχετα με το μέγεθο ε, του αγωνίσματο. Οπότε, άσχετα αν οι υποδομέ είναι μεγάλε ή μικρέ, θα πρέπει να επιλέγονται σε παγκόσμιο επίπεδο και να χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα. Αν συνεχίσουμε αυτόν τον παραλληλισμό με του Ολυμπιακού αγώνε, και αν θέλουμε να έχουμε τοπική επιστροφή, τοπικό όφελος, που δεν είναι μόνο τοπικό αλλά κυρίως τοπικό, από την διοργάνωση μιας και την ε, στέγαση μιας τέτοιας υποδομής, θα πρέπει να κάνουμε ότι με τους Ολυμπιακούς. Συναντήθηκα με τον ε, Ρώσο Υφυπουργό Έρευνα, τον κύριο Γκρούνοφ, και είπε τι εμείς θα πρέπει να πληρώσουμε για να κατασκευάσουμε μια υποδομή στη Ρωσία που θα τη χρησιμοποιήσετε εσείς. Τι κάνατε στο Σότσι, του είπα. Εκεί είναι που διοργανώνετε τους Ολυμπιακούς και άρα κατασκευάζετε το Ολυμπιακό στάδιο, εσείς βάζετε τα χρήματα ε, και έτσι προπονείτε καλύτερα τους αθλητές σας, ε, οι υποδομές θα παραμείνουν σε εσάς και μετά τους Ολυμπιακούς και θα αλλάξετε και το τοπίο και τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής χάρη στη διοργάνωση αυτή που εσείς βέβαια θα χρηματοδοτήσετε. Τέτοιος μηχανισμός προσπαθούμε να μεταφέρθει και στις ερευνητικές υποδομές. Οπότε υπάρχουν και τα διαρθρωτικά κονδύλια. Από πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά, μόνο από τι βόρειε χώρε. Τα διαρθρωτικά κονδύλια δυστυχώ δεν χρησιμοποιούνται με άριστο τρόπο συνήθω. Μακάρι να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα, αυτό θα είναι πρόοδο. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για μακροπρόθεσμη, μακρόπνοη έρευνα και στρατηγικέ μακροπρόθεσμε επενδύσει. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά κονδύλια και να τα αξιοποιήσουμε για να έχουμε πραγματικά μακροπρόθεσμες αλλαγές. Αναφέρθηκε το θέμα της σύνδεσης με τα πανεπιστήμια, με την ανώτατη εκπαίδευση. Οι περισσότεροι χρήστες αυτών των ερευνητικών υποδομών είναι φοιτητέ ή πτυχιούχοι. Αλλά και η κατάρτιση των τεχνικών μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε υπάρχει μια άμεση σύνδεση με την ανώτατη εκπαίδευση. Ευτυχώς όμως αν οι ερευνητικέ αυτές οι υποδομές μπορούν να προσελκύσουν τους καλύτερου, όπως είναι τα Ολυμπιακά στάδια που προσελκύουν τους καλύτερου αθλητές, δεν θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πανεπιστημίων, γιατί συνήθως τα πανεπιστημία, τα πανεπιστήμια οχυρώνονται, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα καλό ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά χωρίς εξυπηρετούν τους άλλους. Για παράδειγμα, όταν κάποιος να δουλεύει στο πανεπιστήμιο δεν θέλει να εξυπηρετήσει τον συνάδελφο, προσπαθεί να απομονωθεί από το συνάδελφο. Ενώ τέτοιε ερευνητικέ υποδομέ στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν και του ε, άλλου. Και αυτό συνιστά μια αλλαγή τη νοοτροπία για του ε, φοιτητέ που χρησιμοποιούν αυτέ τι ερευνητικέ υποδομέ. Και ένα βήμα φυσικά προ τη σύνδεση με τα πανεπιστήμια. Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σας κύριε Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ε, κουνιέται πολύ στην καρέκλα του ο πρόεδρος, φαίνεται να δυσανασχετεί. Κυρία Τόγια, έχουμε εδώ μια άμεση σχέση με ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι ότι οι κανονισμοί, και αυτό το θέμα σχετίζεται και με τα διαρθρωτικά ταμεία, οι κανονισμοί που καταρτίστηκαν για εμπορικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να ισχύουν ούτε για τον αθλητισμό ούτε για την έρευνα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από έναν αθλητή ε, να μας πει, να μας προεξοφλήσει ποιο θα είναι το ρεκόρ του. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε έναν ερευνητή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνάς του. Μπορούμε όμως να του ζητήσουμε να είναι ενθουσιώδης, φιλόδοξοι και να προχωρήσουν πέρα από τους προκατόχους τους. Και με τη φιλοδοξία αυτή θα προωθήσουν και τη γνώση και την τεχνολογία και την οργάνωση. Τώρα, ποια είναι η βέλτιστη οργάνωση. Ευτυχώς στην Ευρώπη δοκιμάσαμε κάποιες οργανώσεις, ε, το CERN, το EMBL. Αυτά τα διακυβερνητικά όργανα, αυτές οι διακυβερνητικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν κάποιες, ε, δημιούργησαν κάποιες υποδομές από τη δεκαετία του 50 και μετά και ήταν πολύ αποτελεσματικά όλα αυτά τα όργανα και έφεραν την Ευρώπη σε ένα πολύ καλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και μάλιστα στηρίχθηκαν περισσότερο στην εμπιστοσύνη και όχι τόσο στο σχολαστικό έλεγχο ή στην μικροδιαχείριση. Γιατί ένας σχολαστικός έλεγχος μπορεί να μετατραπεί σε μικροδιαχείριση. Οπότε το, συμβουλίο, το, το Ινστιτούτο ΕΡΙΚ ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι αποσυνδεδεμένο από του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθω λέει ότι γι' αυτό φταίει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι ο υπέτειο αυτή τη κατάσταση. Το θέμα είναι ότι. Το ξέρω ότι δεν ευσταθεί κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι η υπερβολικό έλεγχο επιφέρει μία καμψία. Και θα πρέπει να δεχτούν περισσότερο ε, ε, το ρίσκο και να εξασφαλίζεται μεγαλύτερος επιστημονικός έλεγχος. Όπως ε, ο έλεγχος που ασκεί η Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για παράδειγμα. Δεν σταματάμε τον αγώνα στη μέση για να δούμε, να ελέγξουμε αν το μέχρι τώρα αποτέλεσμα είναι το σωστό. Τέτοιου είδους ε, ε, ελαστικότητα χρειαζόμαστε. Στην Ιταλία, στη Γερμανία και στην Γαλλία είχαμε διάφορα Ινστιτούτα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία Είχαμε τη Société Civile, που είναι μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα οργάνωση. Ε, στην Ιταλία δεν έχουμε κάτι τέτοιο, είναι πιο άκαμπτα τα πράγματα. Στη Γερμανία επίσης ξέρω ότι υπάρχει μια νομική οντότητα. Στην ε, Μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα φέρουμε στο ΕΡΙΚ και να αξιοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι βέβαια δεν έχουμε ήδη πολλά ΕΡΙΚ, γιατί μόλις τον Αύγουστο, το προηγούμενο Αύγουστο εγκρίθηκε, αλλά τουλάχιστον 10 υποδομές έχουν ξεκινήσει χρησιμοποιώντας τη δομή του ΕΡΙΚ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που δεν έχουμε ακόμη πολλά ΕΡΙΚ. Ελπίζω να ικανοποίησα τις απορίες σας, τουλάχιστον ε, τις πιο συχνές και επίμονες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πληροφορίες, προτάσεις, αρεθίσματα και είμαι σίγουρος πως δεν είναι η τελευταία φορά που σας βλέπουμε γιατί το θέμα βεβαίως μας αφορά όλους και θα μας απασχολήσει οπωσδήποτε τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, τη βοήθειά σας και τελειώσαμε εδώ με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 15. Κοινοτική πολιτική για την καινοτομία σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Να ζητήσω, να δώσω τον λόγο στον κύριο Βίνκλερ, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχετε το σχέδιο έκθεσης. Είναι μια προσπάθεια να ασχοληθούμε με τη μελλοντική κοινοτική πολιτική για την καινοτομία σε περιορισμένο χώρο. Είμαι σίγουρος πως δεν περιέχονται εδώ πέρα τα πάντα όσα σκέφτομαι εγώ αλλά και οι συνάδελφοι βεβαίως γιατί δεν αρκεί ο χώρος αλλά ίσως κάπου με κάποιες ε, τροπολογίες ε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το κείμενο. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους και οδης εισηγητές, αλλά και τους συναδέλφους εκείνους που ήδη κατέθεσαν προτάσεις για το πώς ε, θα γίνει καλύτερο το κείμενο. Για το θέμα τώρα συνέργεια των διαφόρων προγραμμάτων πλαισίου και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει κάποια επικάλυψη με την έκθεση των συναδέλφων Ρόι και Χατζημαρκάκη και του Παλ Ρούμπιχε, κάτι το οποίο εκθέσεις τις οποίες συζητήσαμε και σήμερα το πρωί. Διάβασα επίσης το σχέδιο έκθεσης ε, της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και υπάρχει και εδώ πέρα αρκετή ε, επικάλυψη. Κάποια πράγματα τώρα για τη βάση αυτής της έκθεσης. Η έκθεση βασίζεται στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν από τον Σεπτέμβριο του 2009, επανεξέταση κοινοτικής πολιτικής για την καινοτομία σε έναν απέναντι κόσμο στις 2 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια όπου καταγραφεί η πρόοδος από το 2005 και επίσης αφορά και τις τεχνολογίες κλειδιά έρχεται αυτή η έκθεση σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία αυτή τη στιγμή η Κομισιόν κατανέμει αρμοδιότητες και πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε καθώς ε, έχουμε και το σχετικό νομοθέτημα το οποίο από το Μάρτιο αναβλήθηκε για το καλοκαίρι οπότε εμείς έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε κάποιες, ε, κάποια ρεθίσματα, κάποιες απαιτήσει να αναπτύξουμε στην Κομισιόν για το πώς θα επιτευχθούν οι ουσιαστικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σχεδίου αυτού δράσης. Εγώ θα αναφέρθω τώρα στα σημαντικότερα κατά την άποψή μου σημεία του σχεδίου έκθεσης. Υποθέτω πως και θα το διαπιστώσετε άλλωστε πως η καινοτομία παρουσιάζεται ως το μέσο εκείνο για να αντεποκριθούμε στις κοινωνικές και οικολογικές ε, απαιτήσεις του μέλλοντος ε, και βεβαίως ε, αυτές είναι η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, το πρόβλημα της απασχόλησης και η, δημοκρατική, η δημογραφική με αλλαγή που θα μας απασχολήσει. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια ευρύτατη προσέγγιση για την καινοτομία. Μιλάμε για τεχνολογική αλλά και μη τεχνολογική καινοτομία ειδικά μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει και η κοινωνική καινοτομία να ληφθεί υπόψη, να μετράμε και την κοινωνική και όχι μόνο την οικονομική και οικολογική αξία της καινοτομίας και εδώ πέρα ευχαριστώ τον συνάδελφο την κυρία Καρβάλιο Δεκαστήγιο για το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε συνέπειες όπως η γύρανση της ε, κοινωνίας, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει με τις λεγόμενες τεχνολογίες κλειδιά και τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές όμως πως θα πρέπει να ενισχύσουμε εδώ πέρα τη συνεισφορά μας και βεβαίως να μην ενισχυθούν μόνο οι λεγόμενοι φάροι, οι μεγάλες επιχειρήσεις και πόλη, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που μπορούν να επιτύχουν τεχνική πρόοδο. Οπότε πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι το βασικό μας θέμα εδώ πέρα και του νομοθετήματος περί καινοτομίας. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα η μικρομεσαία επιχείρηση να εφαρμόσει ε, ε, καινοτόμες διαδικασίες, να υπάρξει απλοποίηση της διοίκησης, ε, να μπορέσει να διασφαλίσει καλύτερα την πνευματική της ιδιοκτησία και όλα αυτά. Οπότε έχουμε την πολιτική των πόλων, των clusters και να ενισχύσουμε βέβαια και τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ε, τομείς για να γίνει ακόμη πιο ελκυστική η Ευρώπη. Όλα τα επίπεδα δράσης πρέπει να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία. Σημαντικό είναι επίσης ο προϋπολογισμός της Ένωσης για την καινοτομία να αυξηθεί και να υπάρξει στοχευμένη η προώθηση μέτρων που έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στο μέλλον θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δομές της διοίκησης Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν διπλές ενισχύσεις, αλληλεπικαλύψεις και τα λεφτά και πρέπει να τα εμποδίσουμε όλα αυτά. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαμόρφωση των προγραμμάτων. Το κενό μεταξύ έρευνας και καινοτομίας και ε, διάθεση στην αγορά πρέπει να κλείσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιτρόπων και γενικών διευθύνσεων, κατά το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο με βάση την κατανομή των χαρτοφυλακίων της νέας επιτροπής και βεβαίως πρέπει να έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση και περισσότερη χρηματοδότηση και από τον ιδιωτικό τομέα και από πλευράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και εγγυήσεις βεβαίω μικροπιστώσεις και δάνεια και θα πρέπει να δώσουμε βάση και αυτό έχει σημασία για όλο και περισσότερους συναδέλφους πως ε, συνολικά οι συνθήκες ε, πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθούν, να μην έχουν τόσο γραφειοκρατικό βάρος, να μην έχουν συνέχεια υποχρέωση αναφοράς, έτσι ώστε ο αέρας της καινοτομίας ε, να υπάρξει, να υπάρχει δηλαδή και χώρος να κινηθούν αυτές οι επιχειρήσεις κτλ. Äh, Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα η σκιώδη συγκέντρια κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίγκλερ. Συμφωνώ απόλυτα για με το σχόλιο σα για τις μικρομεσαίες. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και την ε, σημασία τη καινοτομία, κύριε Δίγκλερ. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της καινοτομία και της εμπορευματοποίηση των προϊόντων. Πού βρίσκεται όμως το χάσμα αυτό, μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας ή μεταξύ της καινοτομίας και της θέσης εμπορία μεταξύ της καινοτομίας και της αγοράς δηλαδή. Όπου και αν βρίσκεται πάντως αυτό το κενό, αυτό το χάσμα θα πρέπει να το γεφυρώσουμε και εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Για την καινοτομία δεν θα πρέπει να την περιορίσουμε. Να μην έχω μια συσταλτική ε, άποψη της καινοτομίας. Η καινοτομία χρειάζεται και οριζόντια και κατακόρυφη προσέγγιση και φυσικά απαιτεί συμμετοχή των επιχειρήσεων, των βιομηχανικών κλάδων, των κυβερνήσεων και των πολιτών. Και η συμμετοχή των πολιτών, η συμμετοχή των καταναλωτών είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές παραγωνίζονται και εξοβελίζονται από τη συμμετοχή στην καινοτομία οι καταναλωτές, οι πολίτες. Είναι πολλά τα επίπεδα της ανάμειξης και θα πρέπει να μην αμελήσουμε κανένα από αυτά. Και το ευρωπαϊκό και το κυβερνητικό είναι σημαντικό χρειάζεται και διακυβερνητική και υπερεθνική συνεργασία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιφέρουμε διαρθρωτικές αλλαγέ και να μην μιλούμε μόνο για καινοτομία, αλλά για αηφόρο καινοτομία, γιατί μας ενδιαφέρει μια φιλοπεριβαλλοντική πράσινη οικονομία. Και από αυτή την άποψη η καινοτομία θα πρέπει να προσανατολιστεί στην διαμόρφωση μιας αηφόρου κοινωνίας. Γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το ζητούμενο και χρειαζόμαστε μεταστροφή από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο φιλοπεριβαλλοντικά καύσιμα και φυσικά χρειαζόμαστε και αλλαγή της νοοτροπίας. Η καινοτομία είναι πανταχού παρούσα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ε, σε όλα τα επίπεδα και περιμένω στις συναντήσεις με τους επιτρόπους να επιμείνουμε σε αυτή την αριζόντια προσέγγιση δεν είναι μόνο η έρευνα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην καινοτομία. Υπάρχει η κοινωνική καινοτομία, η καινοτομία της κοινωνίας, ψυχολογική καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία. Δεν υπάρχει μία μόνο καινοτομία. Και σίγουρα δεν είναι μόνο η ερευνητική. Θα πρέπει πάντως να βρεθεί η καινοτομία στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ε, πράσινων, οικολογικών και να βρούμε τους σωστούς εργαζόμενους με τα σωστά προσόντα και δεξιότητες. Γι' αυτό και καλό θα είναι να μην ε, αφήσουμε έξω από τη συζήτηση την παιδεία. Βέβαια δεν έχουμε κοινοτικέ αρμοδιότητες για θέματα παιδείας, αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει κάποιες συστάσεις σε θέματα παιδείας, ώστε να έχουμε ειδικευμένου ε, εργάτες για να μπορέσουν να, ε, να επιτελέσουν σωστά το έργο τους. Μιλήσαμε και για τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σημαντικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν βρίσκονται στο επίκεντρο δυστυχώς. Γιατί είπαμε ότι η καινοτομία και η έρευνα θα πρέπει να προέρχεται κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί έχουν σημαντικό ρόλο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι οι μόνες που έχουν σημαντικό ρόλο. Και οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην καινοτομία. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα σχολιά μου. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον παρακαθήμενο για την γνωμοδότησή του που μας βρίσκει σύμφωνος και χαιρόμαστε για τις παρατηρήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι μόνο οι παραλήπτες αλλά και οι δημιουργοί της καινοτομίας. Και στην ανακοίνωση, για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε τη θέση μας ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς της γνώσης. Αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε πολύ σημαντικά υπόψη. Και νομίζω ότι πολύ σημαντικό σημείο εδώ είναι το θέμα του κοινοτικού διπλώματος Σε Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε δυνατότητα ούτε ισχύ για να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα για πολλού και διάφορου λόγους. Καλό θα ήταν όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφέρει τη γνώμη του για το θέμα αυτό, γιατί αυτό το θέμα είναι ένα σημαντικό θέμα που παραλείπεται δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά ιδιωτικά κονδύλια, γι' αυτό και υστερούμε σε θέματα έρευνας ε, και καινοτομία σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Να βρούμε, στο, αν δεν έχουμε κοινοτικό δίπλωμα ευρυστεχνίας, κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Και να δούμε πού θα αναζητήσουμε αυτές τις αναλλακτικέ λύσεις. Νομίζω ότι αυτά τα δύο σημεία είναι πολύ σημαντικά για την πολιτική ομάδα. Κατά του λοιπού συμφωνούμε με τον εισηγητή και τον συγχαίρουμε για την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντελκαστίγιο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, γιατί όντως συμπλήρωσε θαυμάσια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό και θα παρακαλούσα να το συμπεριλάβει στην έκθεση του κύριου Βίγκλερ. Το θέμα αυτό αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής και τον έλεγχο της εφαρμογής των διαφόρων στόχων. Γιατί πολύ συχνά ακούσαμε προτάσεις, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Δεν έγινε μια παρακολούθηση και έτσι οι ιδέες έμειναν σε θεωρητικό επίπεδο και παρέμειναν στο επίπεδο των αγαθών προθέσεων. Δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Καλό θα ήταν λοιπόν και για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για τις δικές μας, να υπάρξει μια παρακολούθηση και να δούμε πού έγκυται τα κολλήματα και τι δράσεις απαιτούνται για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση, να δούμε σε ποιο βαθμό υλοποιούνται οι στόχοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε κρατικό επίπεδο, όταν πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Νομίζω ότι έτσι θα δοθούν ενάυσματα, αλλά και θα συγκεντρωθούν και πληροφορίες για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, για το θέμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχουν γραφειοκρατικές δυσκολίες που εμποδίζουν αυτή την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί μπορούμε να μιλούμε για το πρόβλημα αυτό, αλλά αν δεν έχουμε δείκτες και στατιστικά στοιχεία που να μας παρουσιάζουν την κατάσταση για να δούμε αν υπάρχει εξέλιξη και μάλιστα με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, γιατί υποκειμενικές απόψεις υπάρχουν πολλές, αλλά πολύ συχνά δεν υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρφωση μιας γνώμης. Επιμένω λοιπόν σε αυτό το θέμα. να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πιο συστηματική χρήση μηχανισμό για τον έλεγχο της υλοποίησης των στόχων. Να δούμε ποιες είναι οι επιδόσεις, ε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, αν τηρούνται και κατά πόσο υλοποιούνται οι στόχοι. Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για την καινοτομία, αλλά και για όλα τα θέματα των πολιτικών μας. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βίνκλερ για την πολύ αξιόλογη εκθεσή του και να υποβάλω πέντε συστάσεις που κατά κάποιο τρόπο καλύπτονται από το έγγραφο. Είπαμε ότι καλό θα ήταν να διευρύνουμε τον ορισμό της καινοτομία. Αναφέρθηκε η κοινωνική καινοτομία, αναφέρθηκε η οργανωτική καινοτομία. Εγώ θα πρόσθετα και την περιφερειακή καινοτομία. Γιατί η επιστήμη είναι οικουμενική, αλλά η καινοτομία μπορεί να έχει περιφερειακή βάση. Χρειαζόμαστε ανοιχτή καινοτομία. Δεν μπορούμε να έχουμε επιστήμη καινοτομία απομονωμένη. Είναι σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη ανοιχτή καινοτομία. Επίσης, ε, περισσότερα κονδύλια για την παιδεία, για την έρευνα και την καινοτομία. Να δημιουργήσουμε πρόσφορα έδαφος για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιωτικά κονδύλια. Επίσης, θα πρέπει να γίνει συντονισμός της καινοτομίας για να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός και τέλος να ληφθεί υπόψη σημαντική πρόκληση όπως είναι ενεργειακός ανεφοδιασμός και ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασμού το θέμα της γύρασης του πληθυσμού, των νέων ε, νόσων, ε, των παλιών νόσων. Υπάρχουν και πολλά θέματα της κοινωνίας που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την έρευνα και την καινοτομία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Για εμένα αυτό το οποίο προέκυψε από τη συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή πως κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συνεχώς ε, παραγνωρίζονται όταν μιλάμε για την ε, καινοτομία, ενώ ξέρουμε πως όλοι οι προμηθευτές είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν και τους περισσότερους φόρους Οπότε νομίζω πως ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε πέρα από τη φορολόγηση στις επιχειρήσεις να βάλουν στην άκρη και ένα κεφάλαιο κινδύνου το οποίο θα διοχετεύσουν στην έρευνα για να μπορέσουν ακριβώς αυτές τις καινοτομίες να τις μετατρέψουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ε, ακριβώς εκεί εμπεριέχει το κίνδυνο, ότι δεν ξέρουμε εάν θα τα προτιμήσουν αυτά οι καταναλωτές, γιατί από εκεί εξαρτάται η επιτυχία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω και νομίζω το ανέφερε σωστά ο συνάδελφος ο κ. Βίγκλερ, πως ε, θα πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση φοροαπαλλαγών και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, κυρίως όταν μιλάμε για επιχειρήσεις ε, νέας ε, τεχνολογίας και θα πρέπει να αναπτύξει νέες ιδέες η Κομισιόν κατά το οποίο δεν ε, μου ενέπνευσε ο κύριος Κόβατς αλλά ελπίζω ο νέος Επίτροπος να σκεφτεί τι θα κάνει για την εσωτερική αγορά στον τομέα της φορολογικής πολιτικής καθώς έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα διπλή φορολόγηση και πάρα πολλά εμπόδια όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό νομίζω είναι σημαντικό ο τομέας ε, της πολιτικής καινοτομίας σε έναν κόσμο που αλλάζει να συνδεθεί και με την νομοθεσία περί μικρών επιχειρήσεων για να εκπληρωθούν οι στόχοι που αναφέρονται εκεί πέρα και καλό θα ήταν η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να κάνει εδώ μία αξιολόγηση αντικτύπου για το αν αυτά τα οποία έχουμε εδώ πέρα επιτάπητος ε, συμφωνούν με το Small Business Act και ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούια. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Σάλφο Βίνκελ για μια ενδιαφέρουσα και πλήρη έκθεση. Δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Εκτιμώ το γεγονός ότι μίλησε για μια πολιτική καινοτομία ευρύ, ευρέως φάσματος ε, γιατί είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη μονάχα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες περιμένουν αυτήν την πράξη με πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες και επίσης το ότι λαμβάνει υπόψη και τομείς ακόμα πιο καινοτόμου, α πούμε μικρο και νάνο ηλεκτρονική. Εκεί ξεκινάει κοινή πολιτική έρευνας ε, και καινοτομίας ε, και πρέπει να δούμε εάν θα στηριχτούν αυτές οι νέε τεχνολογίε. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία όπω α πούμε η ποσοτική καθώς επίση και άλλοι τομείς ε, που μπορεί να φανούν πολύ ενδιαφέροντε τεχνολογίε υγεία επίση, πολύ ενδιαφέρον τομέας. Ε, καθώς επίσης σημαντικές είναι και οι τα πιλωτικά ε, προγράμματα αυτές, δηλαδή οι πιλωτικές ε, πρωτοβουλίες οι οποίες θα δείξουν κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα ή όχι τα, τα προγράμματα. Μπορεί να είναι λίγες αυτές ε, οι πιλωτικές πρωτοβουλίες, αλλά κάποιες έχουν προχωρήσει. Επίσης, ε, εκτιμώ και θέλω να στηρίξω το αίτημα για περισσότερα κονδύλια στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτό μπορεί να ισχύει ε, και για το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, αλλά και για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν καρπούς, αλλά χρειαζόμαστε περαιτέρω κονδύλια και οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι για να υπάρξει ανάπτυξη ή αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη, οπωσδήποτε ε, θα στηριχτεί στην έρευνα και στην καινοτομία και επομένως χρειάζεται και πραγματική στήριξη και όχι μονάχα κάποιες κατευθυντήρες γραμμές. Επίσης, σχετικά με όσα είπε η Συνάχος Πιλάρντε Καστήλιο, συμφωνώ και εγώ ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την νέα νομοθεσία απλώς εκφράζοντας την βούληση της Επιτροπής μας. Ε, τα έχουμε πει, θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία, θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα ε, κάποια στιγμή, ενώ τα έχουμε πει τόσες φορές, θα πρέπει να τα βάλουμε ε, πολύ σαφώς τα, τα σημεία αυτά, γιατί μέχρι τώρα ε, τα εκφράζουμε σαν σημεία κλειδιά ε, μέσα από κανονισμούς, μέσα από εκθέσεις, μέσα από ε, άλλου είδους δραστηριότητες, αλλά τελικά δεν ξέρουμε πού καταλήγουν. Εμείς πρέπει τα σημεία αυτά κλειδιά να τα πούμε σαφώς και να δούμε εάν γίνονται δεκτά ή όχι. Αυτό είναι καλό και για μας, αλλά και για τους ψηφοφόρους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαλός. Από την ΟΚΕ. Ε, euh, euh, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θέλει να έχει πάντα ορθολογική άποψη. Γι' αυτό λοιπόν ε, οργάνωσε ακρόαση για αυτό το θέμα της χειροτομίας και πήγαμε στο IPTS στη Σεβίλη που είναι ακριβώς το κέντρο έρευνας ε, της Κομισιόν και της Επιτροπής που εργάζεται ακριβώς για τις ε, ε, δημοσιονομικές προοπτικές και την καινοτομία και ήρθαμε σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους τομείς και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα. Τα συμπεράσματα θα υποβληθούν την επόμενη εβδομάδα στην αντίστοιχη Επιτροπή της ΟΚΕ. Βεβαίως ε, για μας η καινοτομία πρέπει να είναι και η καινοτομία στις επενδύσεις ε, και η καινοτομία σε κοινωνικές επενδύσεις, ε, η καινοτομία όσον αφορά την διοίκηση, την γραφειοκρατία, αλλά επίσης και τις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες γνωρίζετε ότι και αυτές πρέπει να προωθηθούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταδείξουμε ότι είναι ανόητο, είναι παράλογο λόγο μάλλον ακόμα σήμερα να έχουμε κατακαιρματισμένες ε, πολιτικές όσον αφορά τη βιομηχανία και την τεχνολογία. Η μεγάλη αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν ακριβώς ότι δεν ενέταξε την έρευνα και την ε, ε, καινοτομία σε ένα ευρωπαϊκό πεδίο. Επίσης, μέσα από την ε, σύγκριση ανάμεσα του Small Business Act και αυτά τα προγράμματα καινοτομία ε, Τα συγκρίναμε λοιπόν όπως πρότεινε και ο ε, κύριος Ρουιμπίχ και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία εν μέρη μας εξέπληξαν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις παρουσιάσεις από τρεις γενικές διευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα της ε, καινοτομία. Ε, ήταν στα πλαίσια μια ε, συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδαμε ότι ακόμα και η κάθε μία από τι γενικέ διευθύνσει προσπαθούσε να πει ότι η καινοτομία είναι δικό τη θέμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια καταθμημένη προσέγγιση προ, πρόθεση λοιπόν της ε, καινοτομίας με καλύτερη οργάνωση, με καλύτερες υποδομές αλλά και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι και πρέπει να έχουμε μάλιστα ευρωπαϊκή φιλοδοξία όσον αφορά την καινοτομία και να προχωρήσουμε με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαλός. ευχαριστώ πάρα πολύ και θετικό είναι ότι είστε και παρόν εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα τον λόγο στην Κομισιόν, ο κύριος Ντρόλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνεισφέρω και εγώ θεωρούμε πως μας ενθαρρύνει στο περαιτέρω έργο μας. Αυτή η έκθεση να δίνει σαφείς αφετηρίες για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Αυτά που αναφέρθηκαν συζήτηση, απλοποίηση, κατάργηση γραφειοκρατίας, βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια ευρεία προσέγγιση, είναι σημαντική η έρευνα για να δημιουργηθεί γνώση από την οποία θα προκύψει η καινοτομία, αλλά είναι μία συνεισφορά αυτή. Χρειαζόμαστε τον καταναλωτή, τον χρήστη, και να απευθυνθούμε στους μεγάλους κοινωνικούς στόχους και αυτό σημαίνει πως πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα, τα μέρη, τα ενδιαφερόμενα. Ο κύριος Βίγκλερ είπε πως πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ πέρα όλα τα επίπεδα της δράσης και πράγματι πρέπει να, εξετάσουμε πώς θα το επιτύχουμε αυτό. γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παίκτη μόνο εδώ πέρα. Εάν δούμε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, βεβαίως είμαστε πολύ ισχυροί, αλλά εάν μιλήσουμε για την εκπαίδευση, που είναι πολύ ουσιαστική, έχουμε μικρό ρόλο να παίξουμε και εκεί πέρα έχουν να παίξουν ρόλο τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε σε αρχές οι οποίες ε, θα κατευθύνουν το ευρωπαϊκό σύστημα καινοτομία για να υπάρξει μια συμφωνία εν μέσω όλης αυτής της ποικιλία ε, των δράσεων. Αυτά από εμά. Συμφωνώ πλήρως με την παρατήρηση πως χρειαζόμαστε στόχους, δείκτες, μετρήσιμους, με τους οποίους ε, θα πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε αν επιτύχαμε τους στόχους μας. Αυτό λείπει δεν είναι σύμπτωση γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτύξουμε δείκτες για την πρόοδο της καινοτομίας και να μετρήσουμε κάτι. Αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας για τη μελλοντική στρατηγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτά. Νομίζω και σήμερα. Ή κύριε Βίνκλερ, ε, θέλετε πάλι το λόγο. 2 μέχρι τις 2 Μαρτίου για τις ε, τροπολογίες είναι η προθεσμία, οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 16. Mobilisierung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Übergangs zu einer κινητοποίηση των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση μετάβαση προ μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα. Η κυρία Τόγια είναι η συγγήτρια η οποία έχει τον λόγο πρώτη. Για να μας πει τι έχει να μας πει και μετά οι συνάδελφοι. Η κυρία Τόγια έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο έκθεσης, όπως και εσείς είπατε, αναφέρεται στην χρήση των TIC, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια ενεργειακά αποδοτικότερη η ε, οικονομία και ακριβώς να μελετήσει τον ρόλο ε, που μπορούν να έχουν ε, τα ITC προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μία ανακοίνωση του προηγούμενου Μαρτίου, καθώς επίσης και μία σύσταση στο, του φθινοπόρου του 2009, ε, που ε, περιγράφουν τις δυνατότητες του τομέα ε, να ε, μπορέσει ακριβώς μέσα από τις δικές του δυνατότητες με καλύτερη οργάνωση εργασίας, με καλύτερη χρήση του προϊόντος ε, της εργασίας τους ε, να γίνουν πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και όσον αφορά και τις ίδιες τις δραστηριότητες καθώς επίσης και την σημαντική συμβολή αυτού του τομέα σε άλλους μέσα από τις μεταφορές, μέσα από, τη, από προγράμματα στέγασης, έτσι ώστε να έχουμε αφενός εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Ανοίγουν ευρύτατα πεδία δράσης που επανειλημμένα έχουν συζητήσει και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και ε, ε, βεβαίω αναφέρονται μία σειρά ε, προκλήσεων και διακυβευμάτων όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πιστεύουμε ότι το κοινοβούλιο, και το Κοινοβούλιο γενικώ πιστεύει ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι πιο δεσμευτικοί έτσι ώστε να περάσουμε σε μία πραγματικά ενεργειακά αποδοτικότερη οικονομία και πιο αποτελεσματική μάλιστα ε, η οικονομία. Ε, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και την ε, γραμματεία μας αλλά και τις υπηρεσίες της Επιτροπής με τους οποίους συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά στη διάρκεια της προετοιμασίας. Βεβαίως δεν μπορέσαμε να δεν είχαμε τον χρόνο να ενσωματώσουμε στην έκθεση όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν την προηγούμενη φορά που συζητήθηκε το θέμα. Υπόσχομαι όμως ότι και μέσω τροπολογιών Λοιπόν θα προσπαθήσω να αντικατοπτρίσω στο κείμενο όλες αυτές τις ε, απόψεις. Ήδη από τα πρώτα σημεία της έκθεσης ε, γίνεται σαφές ε, ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εδώ γίνεται αναφορά στο 2010, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε ε, έτσι ώστε μέχρι τότε να υπάρξουν συγκεκριμένες συστάσεις ε, οι οποίες θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των πιλωτικών ε, προγραμμάτων. Επίσης και την δυνατότητα της ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Να δώσουμε ε, λοιπόν την δυνατότητα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών καθώς επίσης και άλλων τεχνολογιών που είναι απλές, εύχριστες, ε, οι οποίες ε, μπορούν άμεσα να διατεθούν στους καταναλωτές έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογικότερη χρήση και κατανάλωση ενέργειας, έτσι ώστε να ρυθμιστεί αυτή η κατανάλωση ενέργειας και έτσι ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και οι καταναλωτές σε αυτήν την προσπάθεια εξοικονόμησης ε, και καλύτερης χρήσης ε, ενέργειας. Μία αμφίδρομη λοιπόν ε, σχέση που θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης γνώσης του ποσοστού κατανάλωσης αλλά και του τρόπου κατανάλωσης. Σήμερα το πρωί για ένα πάρα πολύ σημαντικό φόρουμ για αυτό το σημαντικό θέμα και μάλιστα ε, ε, το σημαντικό θέμα της, ε, της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για την καλύτερη και ενεργειακά αποδοτικότερη η οικονομία και μάλιστα θα υπάρξει και μία έκθεση έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το εργαλείο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας να γίνει ένα σημαντικό κλειδί επικοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν πιλωτικά προγράμματα, υπάρχουν οι τεχνολογίες και επομένως ε, θα πρέπει να διαχυθούν οι τεχνολογίες αυτές. Ένα άλλο θέμα, ουσιώδες κατά την άποψή μας, ε, το οποίο ε, απέρασε και από την διαβούλευση που πρόθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά, ε, επαφές ε, με εμπειρογνώμονες, ε, με χρήστες αλλά και με operators του τομέα αυτού. Στα πλαίσια λέγω της διαβούλευσης αυτής έγινε σαφές ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με όλους αυτούς τους φορείς και να εκπονηθεί μεθοδολογία βάσει της οποίας θα οδηγηθούμε σε κοινέ διαδικασίες και σε κοινά ε, πρότυπα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξουν στάνταρ διαδικασίες όσον αφορά την χρήση αυτών των έξυπνων μετρητών που ανέφερα και προηγουμένως ε, και άλλων τέτοιων εργαλείων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν έχουμε κοινά, ε, ε, κοινές μεθόδους ε, μέτρησης, κοινές διαδικασίες, κοινά χρονικά περιθώρια. Αυτές είναι λοιπόν προτάσεις οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να ξαναδούμε εάν χρονικά μπορούν τα κράτη να ανταποκριθούν σε αυτές ή αν θα πρέπει να επιμηκύνομαι της προθεσμίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι Μέχρι τώρα έχουμε σποραδικές και κατακαιρματισμένες ε, εμπειρίες ενώ εμείς και μεθοδολογίες ενώ εμείς θέλουμε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα και μια ενιαία μεθοδολογία. Αυτά είναι τα σημεία που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά. Εκτιμούμε επίσης την πρόταση της Κομισιόν να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, μια task force για τα έξυπνα συστήματα μετρητών και βεβαίως ε, μας ε, ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η προώθηση των, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας, δεσμευτικές λοιπόν, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί κάποιων διαδικασιών. Ε, βεβαίως ε, εδώ στην έκθεση ε, αναφέρω το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το ποιο θα είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορούμε να το δούμε όλοι μαζί, να δούμε ε, τι θα πρέπει να αποφασίσει η Κομισιόν, τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν, τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, ε, πόσο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να εμπλέξουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, κυρίως και τις ενδιαφερόμενες ε, επιχειρήσεις, ε, δημόσια διοίκηση των ε, κρατών μελών που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί πρέπει να ξέρουμε τι, πώς χρησιμοποιούν τα κρατημέλη, πώς χρησιμοποιεί η διοίκηση των κρατών μελών αυτές τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στον τομέα της υγείας και σε ένα σωρό άλλους τομείς. Ένας οδικός χάρτης λοιπόν, ένα φύλλο μάλλον που θα είναι δεσμευτικός και όποιος αποφασίσει να ακολουθήσει το φύλλο πορείας να έχει ήδη ε, μία προδιαγραμμένη πορεία που θα τον ε, βοηθήσει. Μίλησα, εγώ αναφέρθηκα σε κάποιους ε, τομείς βιομηχανικούς και τον ρόλο των κρατών μελών, αλλά υπάρχει το μεγάλο ζήτημα των μεγάλων πόλεων που βρίσκουμε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλες τις χώρες μέλη υπάρχουν μεγάλες και εκεί το ζήτημα της διοίκησης είναι πιο σοβαρό. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της θέρμανσης, πώς αντιμετωπίζονται ε, πολλά ζητήματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Φαίνονται πολύ λίγα, πολύ μικρά αυτά. Όταν κανείς δει ε, ένα πρόγραμμα ας πούμε ενεργειακής αποδοτικότητας ε, διαπιστώνει ότι απαρτίζεται από πολλά μικρά πράγματα τα οποία όμως μπορούν στην σωστή τους εφαρμογή να ε, οδηγήσουν όπως ας πούμε οι έξυπνοι μετρητές σε μείωση ακόμα και 10% της κατανάλωσης ενέργειας και επομένως μέσα από αυτά τα μικρά πράγματα όταν αυτά τα μικρά πράγματα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς, τότε πραγματικά μπορεί να οδηγήσουν σε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πρόκειται για βήματα τα οποία ε, είναι μικρά, αλλά μας οδηγούν σε μια μακρά πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λάμπερτς. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστούμε και την κυρία Τόγια. Ευχαριστούμε και την κυρία Τόγια για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι υπήρξε εξέλιξη στην προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλό είναι να το τονίζουμε. Τελευταία μιλούσαμε για διοξίδιο του άνθρακα και ενεργειακή αποδοτικότητα. Νομίζω ότι το θέμα που μας ενδιαφέρει είναι κάπως ευρύτερο. Είναι η αποδοτικότητα των πόρων μας γενικότερα. Και αυτό τον έφερε και ο πρόεδρος Μπαρόζο στην Ολομέλεια. Μίλησε για την ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων μας και όχι μόνο τη ενέργειας ειδικά. Και μια συμβουλή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της ήταν να υιοθετήσει αυτή την πιο ευρύτερη θεώρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, της αποτελεσματικότητας των πόρων και όχι μόνο της ενεργειακής ή της, του άνθρακα. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι αυτοί οι ευφυείς μετρητές, το smart metering που αναφέρει και η κυρία Τόγια. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέμε. Όχι ότι δεν χρειαζόμαστε όλο και μεγαλύτερη μετάβαση προς τους ευφύς μετρητές, αλλά με τους ευφύς μετρητές μπορεί να έχουμε στα κροδάχτυλά μας ε, την ευφύα, αλλά το υπόλοιπο νευρικό σύστημα δεν ακολουθεί αυτή την πρόοδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ίδια η ραχοκοκαλιά της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη να, να, είναι πρώτα, να γίνει πρώτα ολοκληρωμένη, ενοποιημένη και μετά να γίνει φύση και να μην προσπαθούμε να ξεκινήσουμε από το τέλος, να κάνουμε τα, τις απολύξεις της μόνο της νευρικές έξυπνες ενώ το υπόλοιπο νευρικό σύστημα. Είπαμε ότι οι ευφύες μετρητές μπορούν να συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10% αλλά υπό όρους. Αν έχουμε έξυπνους μετρητές αλλά οι ηλεκτρικέ οικιακέ συσκευέ δεν είναι αντίστοιχα ευφύης. Δεν μπορούμε να δρέψουμε του καρπού αυτή τη εξοικονόμηση. Πρέπει οι έξυπνοι μετρητέ να συνδυαστούν με ευφυεί οικιακέ συσκευέ, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Και ναι, μεν οι έξυπνοι μετρητέ θα χρειαστούν κάποια στιγμή, αλλά να επιταχύνουμε τη χρήση του. Να μην προσπαθήσουμε να τρέξουμε όταν δεν μπορούμε ακόμα να περπατήσουμε. Όποιο βιάζεται σκοντάφτει, γιατί το κόστος ε, χρήσης των ε, εφιών μετρητών είναι τεράστιο, αστρονομικό. Και δεδομένων των ε, επενδυτικών ικανοτήτων των δημόσιων και των ιδιωτικών, αλλά και της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, προτιμώ να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Να μην ζητάμε κάτι περισσότερο από τις δυνατότητε μας. Και νομίζω αυτή τη στιγμή οι έξυπνοι μετρητέ είναι υπερβολικά φιλόδοξοι. Επίσης το θέμα της πρόσβασης είναι πολύ σημαντικό, γιατί και το θέμα της ασφάλειας του καταναλωτή μας ενδιαφέρει. Ιδιαίτερα για τους πιο επισφαλείς τελικούς χρήστες. Να μην χρησιμοποιηθεί αυτός ο δόριο ύπος για, το... για να αποκαρδιωθεί ο κόσμος από τη χρήση του ηλεκτρισμού. Οπότε θα έλεγα να μην υπερβάλλουμε στην ανάγκη των ε, έξυπνων μετρητών, να υπερτονίσουμε την ανάγκη χρήσης εφιούς δικτύου. Τώρα για τις εκπομπές του του άνθρακα. Σίγουρα η ενέργεια είναι ένα τμήμα του περιορισμού των εκπομπών, αλλά και η κινητικότητα είναι το άλλο σκέλος, η άλλη όψη. Και εκεί οι τεχνολογίες πληροφορίε και επικοινωνίες θα μας χρησιμεύσουν. Αν θέλουμε οι τελικοί χρήστες να πληρώνουν ανά χιλιόμετρο, άσχετα χρησιμοποιούν το σιδηρόδρομο, το λεωφορείο, ποδήλατο ή γιοταχή. Από τη που χρησιμοποιούν τις υποδομές, χρειαζόμαστε να προσφύγουμε περισσότερο στη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Το θέμα της έξυπνης κινητικότητας είναι επίσης πολύ σημαντικό και η ιδέα του «pay as you go». Και άλλο πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι το θέμα των τροφίμων, γιατί φαίνεται ότι κατασπαταλούμε πάνω από τη μισή παραγωγή τροφίμων που παράγουμε. Ενώ σε αναπτυσσόμενες χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες είναι λιγότερο από 20% η σπατάλη αυτή. Και θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην έξυπνη κατανάλωση και εκεί οι τεχνολογίες ε, επικοινωνίας και πληροφορίες θα παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί τα τρόφιμα που πετάμε κυρίως είναι τα νοπά που έχουν πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αλλά με αυτή τη λογική δυστυχώς ε, καταστρέφουμε και πετάμε φαγητό που θα μπορούσαμε κάλλιστα, τρόφιμα που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα καταναλώσουμε. Οπότε χρειαζόμαστε και μία έξυπνη ε, α, αλυσίδα για τα νοπά τρόφιμα. Ήδη γίνονται κάποια πειράματα αυτή τη στιγμή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα αυτό. Να μην το ξεχνούμε λοιπόν. Άλλωστε όλη η επιστημιστική αλυσίδα είναι 30 με 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είναι υπεύθυνη για μεγάλη παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Αν πιστεύουμε ότι η αποτελεσματικότητα των πόρων ή ακόμη και η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο περιορισμό του διοξιδίου του άνθρακα αποτελεί επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις εκθέσεις μας, αλλά και σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Στο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, για παράδειγμα, στα αναπτυξιακά ταμεία, στις περιφερειακές πολιτικές, στην γεωργική πολιτική, όλα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως προτεραιότητα αυτή την εξοικονόμηση, την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας των πόρων. Και αυτό θα πρέπει να τονιστεί και στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάπου περιλαμβάνεται σε εκθέσεις, αλλά θα πρέπει να το δώσουμε πιο περίοπτη θέση και να είναι ορατή αυτή η προτεραιότητα σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάριτς. Thank you very much. I would uh, uh, Ήθελα και εγώ να πω ευχαριστώ στην κυρία Τόια το πρώτο σχέδιο εκθεση. Δύο σχόλια. Τρία. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με το θέμα της τυποποίησης. Για να ορίσουμε τι είναι ο έξυπνος μετρητής. Αυτό μάλλον εννοείται στο 15. Δύο ερωτήσεις έχω. Σημείο 9. Συνιστάται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή των οδηγιών περί ενεργειακή απόδοσης για να συμπεριληφθούν και τα κτίρια διαστάσεων μικροτέρων των προβλεπομένων. Ε, έχουμε ξεφύγει λίγο. Γιατί δηλαδή, το να έχουμε έξυπνο μετρητή σε ένα μικρό σπίτι δεν το κάνει πιο αποτελεσματικό εάν δεν έχει καλή μόνωση. Το να έχει ένα κομπιουτεράκι που σου λέει πώ χάνει τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό, απλά θα ξέρει ε, που ξοδεύει τα λεφτά σου αλλά δεν θα βελτιώσει τίποτα. Και ίσως να μπορεί να κάνεις και τίποτα βραχυπρόθεσμα. Οπότε, θα έλεγα εγώ να ξεκινήσουμε στα δημόσια κτίρια και τα μικρότερα κτίρια το βλέπουμε μετά. Είναι σημαντικό, αλλά όπως είπε ο κ. Λάμπερτς, ε, το, το αυγό και η κότα. Ε. Να ξεκινήσουμε από αυτά μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Σημείο 16. Καλεί την Επιτροπή να καταρτήσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από όλοι τομείς του που και όλα τα κράτη-μέρη κτλ. κτλ. Εγώ όταν ακούω δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σκέφτομαι κόστος. Τι λέμε εδώ πέρα. Δηλαδή θα αναγκάσουμε μεγάλες εταιρείες να φύγουν οι σερβερ εκτός Ευρώπης σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Πού είναι δυνατόν. Καταλαβαίνω το νόημα των όσων λέτε. Εντάξει πρέπει να έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά ταυτόχρονα Δηλαδή όταν λέμε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι το κόστος για ευρωπαϊκές θέσει εργασία και τι σημαίνει αυτό μακροπρόθεσμα. Για να συνοψίσω. Να χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο είπε ο κ. Λάμπερτς. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Και αφού γίνει αυτό, α δούμε τι θα κάνουμε μετά. Ευχαριστώ, Ρόντε. και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Τρόια. Ε, πράγματι παρουσίασε σε μια κλειδιά και έκανε μια σημαντική παρουσίαση. Εγώ συμφωνώ με το βάρος που δίνεται στην ε, TPA για τα κοινά πρότυπα, τους έξυπνους μετρητές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πράγματι, εκεί πέρα μπορούν να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα στο πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Αυτό το λέει και η Κομισιόν άλλωστε. Εγώ θα καταθέσω λίγες τροπολογίες, κάποιες για διευκρίνηση, κάποιες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ, τα ΦΠΕ. Μία ερώτηση έχω, ίσως και σύσταση γιατί δεν ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις ε, για δεσμευτικούς στόχους ε, για ενεργειακή αποτελεσματικότητα στον τομέα της ε, ΤΑΦΙΕ. Μας λένε πως όταν έχουμε δεσμευτικούς στόχους, η εμπειρία μας το λέει αυτό, και χρονοδιάγραμμα, οι αγορές όχι μόνο θα επιτύχουν τους στόχους, αλλά συχνά θα τους ξεπεράσουν και όλες. Οπότε όταν η Κομισιόν μας λέει πως τα έξυπνα μέτρα μετρητές μπορούν να εξοικονομήσουν 10% και τα ΦΕ μέχρι 17% από εκπομπέ κτηρίων και 27% από, από τις μεταφορές. Ας γίνουν αυτοί οι αριθμοί στόχοι. Και έτσι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί βεβαίω οι αγορές ακολουθούν τους πρωτοπόρους. κυρία Ρόλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία ε, Τόγια για την εξαιρετική δουλειά της. Συμφωνώ μαζί της ε, όσον αφορά την σημασία των μικρών έξυπνων μετρητών. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Ε, ας μιλήσουμε πρώτα για την οδηγία ενεργειακής αποδοτικότητας των ε, κτίριων. Νομίζω ότι την ξεπεράστηκε από τα γεγονότα γιατί ε, έγινε η αναδιατύπωση της οδηγίας του προηγούμενο Δεκέμβριο και το κατόφλι ήδη έχει κατεβεί στα 50 τετραγωνικά ε, και επίσης ε, έχουμε προωθημένες αιτήσει όσον αφορά την, την καταγραφή της ενεργικής αποδοτικότητας των κτηρίων. Επομένως θα πρέπει να προσαρμοστούμε του ή στην αναδιατύπωση της οδηγία του Δεκεμβρίου. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Λάμπερτς, γιατί πιστεύω ότι οι μικροί μετρητές είναι απόλυτα απαραίτητοι έτσι ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται η τεχνολογία Περάσαμε επίσης νομοθεσίες ε, όσον αφορά τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Πώς είναι δυνατόν οι καταναλωτές να έχουν μία επαφή, να έχουν μία γνώση της ε, κατανάλωσης ενέργειας, εάν δεν έχουν αυτούς τους μικρούς μετρητές, χάνουν την αίσθηση, ξεχνούν ότι ε, καταναλώνουν ενέργεια. Επίσης ε, το θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων προχωράει ε, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι και για τους μικρούς έξυπνους μετρητές μπορεί κανείς να έχει μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία άμεση ε, με τις εταιρείε ε, ηλεκτρισμού και επομένως ε, να μειωθεί και η κατανάλωση, κυρίως δεν αν συνδυαστεί και με νυχτερινή κατανάλωση, να έχουμε πραγματικά εξοικονόμηση ενέργειας. Όσον αφορά τώρα τα κοινά πρότυπα ή τις προδιαγραφές, οι προδιαγραφές είναι ένας μόνο τεχνικός όρος και ενδεχομένως ε, μπορεί κανείς ε, να αναφερθεί ενδεχομένως σε ε, ελάχιστες λειτουργίες. Γιατί γίνεται σαφές ότι κάποιες εταιρείες δεν ενδιαφέρονται τελικά σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους καταναλωτές, δηλαδή η ψηφιακή οθόνη των ε, των μετρητών. Δηλαδή τους ενδιαφέρει εκείνοι σαν εταιρείε να μπορούν να ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας αλλά όχι και οι καταναλωτές να έχουν την ίδια δυνατότητα. Επομένως θα πρέπει οι μετρητές αυτοί να ε, λειτουργούν και να μετρούν την ενέργεια και στην πηγή τροφοδοσίας αλλά και στην, στην κατανάλωση. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Μπάρα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια γιατί πραγματικά είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση. Χαιρόμαστε για την, ανα... την ε, έμφαση που δίνει η έκθεση στην καταμέτρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Χρειαζόμαστε κάποιους κοινέ μεθόδους, γιατί πώς αλλιώς θα συγκρίνουμε ε, την αποτελεσματικότητα των διαφόρων τεχνικών ε, εξοικονόμηση ενέργειας, διαφορέ τεχνικές, διάφορε μεθόδου που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Αν δεν έχουμε κοινέ ε, μεθόδους μέτρησης, πώς θα κάνουμε και τη σύγκριση. Αλλά δυστυχώς χρειαζόμαστε καιρό για να αναπτύξουμε μεθοδολογίες και να καταλήγουμε σε κοινέ μετρήσεις της αποδοτικότητα. Οι ΤΠΕ αναπτύσσονται με ηλικιώδη ρυθμό και μέχρι το 2020 τριπλασιαστεί το αποτύπωμά τους. Και από αυτήν την άποψη ο τομέας ε, των τεχνολογιών πληροφορίες και επικοινωνίας χρειάζεται κάποιες ε, τυποποιημένες μεθοδολογίες και φυσικά να μειώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και για να το κάνει θα πρέπει να υιοθετήσει κάποιες ε, τυποποιημένες μεθόδους μέτρησης για να μπορέσει να καταμετρήσει τα αποτελέσματα των προσπαθειών της. Και αυτό ίσως θα μπορούσε να διευκρινιστεί καλύτερα στην έκθεση. Mm. Τέλος, για τους έξυπνους μετρητές έγινε εκτενή συζήτηση και ήδη υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι στην ε, οδηγία για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Υπάρχουν διορίες ε, για τον οδικό χάρτη αυτών των έξυπνων μετρητών. Οπότε, όπως είπατε πολλοί από εσά στη συζήτηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινό ορισμός για το τι εστί και τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ο έξυπνος μετρητής. Γι' αυτό και υποβάλαμε σύσταση. καλώντας τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στις κοινέ λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί ένας έξυπνος μετρητής. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κυρία Μπάρα για τις πληροφορίες σας αυτές. Οπότε τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. 2 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Κυρία Τόια λοιπόν, παρακαλώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ε, συνέβαλαν στην ε, συζήτηση και να πω επίσης ότι φαντάζομαι ότι το καταλάβατε άλλωστε ότι από την, κατά την άποψή μου όταν ε, παρουσιάζεται ένα προσχέδιο έκθεσης θα πρέπει να είναι ε, κάπως ανοιχτό γιατί δεν έχει έννοια να εμφανίσει μια, ένα προσχέδιο έκθεση ο εισηγητής όπου θα είναι απολύτως αποφασισμένος για όλα τα, τις λεπτομέρειες. Να πω επίσης στον συνάδελφο ο οποίος δεν είναι εδώ πια ότι το, σύστημα, το, ότι το θέμα, το πρόβλημα του κόστους βεβαίως μας ενδιαφέρει Φυσικά ε, σε, οποιοδήποτε, ε, σε οποιοδήποτε πρόταση θα πρέπει να υπάρξει και υπολογισμός κόστους, ευθύπτωσης κτλ. Αλλά πιστεύω ότι μερικές φορές ε, το να ακολουθήσει κανείς ε, ε, μία κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει κάποιο επιπλέον κόστος, αλλά μπορεί να ανοίξει και νέες οδούς στην βιομηχανία. Και βεβαίως κανείς μας δεν θέλει να κάνει κάτι το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσον αφορά τις προδιαγραφές, ε, τα πρότυπα, ναι, ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες ελάχιστες ε, κοινέ αρχές, όπως είπε και η Φιώνα Χολ. Επίσης, ε, βλέποντας ε, ε, αυτό που έγραφε η σύσταση, το οποίο δεν ανέφερα εδώ, γιατί θα ήθελα να εμβαθύνω λίγο στο θέμα αυτό με τους συναδέλφους, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα διαβουλεύσεων και συμφωνιών με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, στους οποίους ε, ζητά σχεδόν να εκπονήσουν επιστολή συστάσεων ε, και προθέσεων. Και εγώ αναφέρθηκα σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα γίνει δεσμευτικό αφού έχει προηγηθεί βεβαίως συζήτηση, διαβούλευση με τους operators του τομέα. και επομένως ε, κάτι το οποίο θα είναι ε, δεσμευτικό αλλά θα έχει αποτελέσει αντικείμενο πρώτερης συνένεσης. Θα είναι κάτι θελημένο δηλαδή, ε, όχι κάτι που θα επιβληθεί. και σας υπόσχομαι ότι οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη όσα ακούστηκαν σήμερα εδώ από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας είπα πότε είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, οπότε τελειώσαμε και με αυτό. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης χρηματοδοτική συνδρομή της κοινότητας για τον παροπλισμό των μονάδων 1 4 του πυρηνικού σταθμού Κόσλο Ντούι. Θα μιλήσω σιγά σιγά γιατί δεν βλέπω την συνάδελφο, την κυρία εισηγήτρια. Κάνουμε ένα διαλυματάκι, δύο λεπτάκια, μέχρι να έρθει η κυρία Χάρμς εδώ πέρα. Να μου λένε ότι έρχεται. One minute. We wait. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Inhalt habe ich gesagt. Kosludui, Finanzhilfe. Richterstatterin ist die Kollegin. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Κοσλοντούι. κυρία Χάρμς θα, θα περιμένουμε λίγο να, να ανασάνει, να ανοίξει το μικρόφωνο και μετά έχει τον λόγο. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αξιολο... αφορά την αξιολόγηση μιας πρότασης Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της ε, απέτησης ε, της... Ε, που προέκυψε στη Βουλγαρία για το ότι σύμφωνα με την συνθήκη προσχώρησης ε, της Βουλγαρίας, η μονάδα 1, 2 και μετά η 3 και 4 θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο και θα συζητήσουμε τώρα το ύψος ε, των ποσών που θα διατεθούν μέχρι το 2013 στη Βουλγαρία. Και κατά την άποψή μου ε, να δούμε και τις προτάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν για την χρήση αυτών των μέσων. Αναφέρω τώρα κάποια σημαντικά νούμερα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε με τις ε, διαβουλεύσεις αυτές. Έχουμε τα 300 εκατομμύρια ευρώ που προτείνει η Κομισιόν ως συνεισφορά της κοινότητας για να σταματήσει η λειτουργία του Κοσλοντούι. Εάν χρηματοδοτηθούν ε, και αυτά έχουμε φτάσει στα 860 σχεδόν, συνολικά σχεδόν όλα από τον κοινοτικό προπολογισμό που θα έχουν πάει στη Βουλγαρία. Με την πρόταση που εξετάζουμε τώρα, το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για τα τελευταία 300 από αυτά τα 860 εκατομμύρια τα οποία κατά βάση θα πάνε σε δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός που προτείνει η Κομισιόν, τον υποστηρίζω εγώ, 180 εκατομμύρια να πάνε δηλαδή για να εγγυηθούμε πως ε, η μονάδα 3 και 4 όπως και η 1 και 2 άλλωστε του Κοσλοντούι θα παροπλιστούν όντως με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να ξαναλειτουργήσουν, κάτι το οποίο είχε συμφωνήσει η Κομισιόν για το Κοσλόντου, Επιπλέον, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να επανεξεταστεί το τι θα γίνει μετά τον παροπλισμό με τα πυρηνικά απόβλητα. Τι γίνεται δηλαδή με αυτά που έχουν παραχθεί από τη λειτουργία. Δεν είναι απλό να έχουμε μία εικόνα της διάθεσης ε, των αποβλήτων από πλευράς ε, Βουλγαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής για τον προγραμματισμό ενδιάμεσης αποθήκευσης για τα υψηλώς ραδιενεργά και ε, σχάσιμα υλικά είναι πως δεν υπάρχει κάποια πρόληψη και κάποιος προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός περιορίζεται στην εξαγωγή, στην ε, επανεξαγωγή θα έλεγε κανείς, προς Ρωσία και από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι μάλλον ανοιχτό το ζήτημα θα έλεγα. Και όπως επίσης ανοιχτό είναι το πότε, πώς και αν θα υπάρξει τελική αποθήκευση στην ε, Βουλγαρία. Επίσης, η πρότασή μου για την περαιτέρω χρησιμοποίηση αυτών των 120 εκατομμυρίων της μη, του μη παροπλισμού θα πρέπει να πάνε κατά την άποψή μου με τον όρο του να μην υπάρξει επεξεργασία στην Ρωσία αλλά να υπάρξει για τη Βουλγαρία να υπάρξει μια λογική αποθήκευση και επεξεργασία στη Βουλγαρία. Με αυτά τα 120 εκατομμύρια νομίζω θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για την ασφάλεια στην Βουλγαρία και μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα στη Βουλγαρία από το να πάνε αυτά τα 120 εκατομμύρια και να πέσουν και αυτά ε, σε αυτή την κατεύθυνση και να μην πάνε σε έργα ενεργειακής αποτελεσματικότητας και άλλα τέτοια παρόμοια. Επιπλέον θεωρώ πως αυτά τα 120 εκατομμύρια Εάν χρησιμοποιηθούν εδώ ή εκεί για ανανεώσιμες ε, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα δεν θα αλλάξουν τίποτα. Δεν πάει η βουλγαρική κατεύθυνση σε αηφόρο, η βουλγαρική κυβέρνηση σε αηφόρο κατεύθυνση γιατί οι Βούλγαροι επιμένουν να χρησιμοποιούν ατομική ενέργεια. Γι' αυτό θεωρώ για λόγους ασφάλειας ε, πως είναι καλύτερο να αναπτυχθεί μια στρατηγική ε, διάθεση των αποβλήτων. Αυτή είναι η διαφορά η ουσιαστική με την πρόταση της Κομισιόν. Το έχουμε σκεφτεί επί μακρόν. Θεωρούμε πως επειδή ο παροπλισμός του Κοσλοντού ιετιολογήθηκε με την περισσότερη ασφάλεια θεωρούμε πως ε, θα πρέπει να προσανατολιστούμε πρώτα απ' όλα στην πυρηνική ασφάλεια στη χρήση αυτών των κονδυλίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελε κάποιος από τους σκιώδεις ηγητές να λάβει τον λόγο ή κάποιος άλλος ε, και ως καθήνα. Uh, Ευχαριστώ. Πολύ καλή έκθεση της κυρίας Χάρμς και βρήθη καλών ιδεών γιατί θέτει μερικά γενικά ζητήματα για την πυρηνική ασφάλεια και για το μέλλον της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Τη συγχαίρω για την έκθεσή της. Επανέρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο θέμα για τον παραπλησμό του Κοσλοντούι. Πρωταρχικός στόχος της έκθεσης αυτής είναι να επιλύσει ένα συγκεκριμένο θέμα και να εξασφαλίσει συνθήκες ε, ελεύθερου ανταγωνισμού και θεμητού ανταγωνισμού για τις, χώρες που, για τις τρεις χώρες που έπρεπε να κλείσουν τα πυρηνικά τους εργοστάσια, τη Λιθουανία δηλαδή, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία και για αυτή τη συγκεκριμένη, με αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση εξασφαλίστηκε η μεταχείριση της Βουλγαρίας με τη Σλοβακία και τη Λιθουανία. Στόχος επίση του προγράμματος αυτού ήταν να βοηθήσει τη Βουλγαρία να αναλάβει αυτό το δυσβάσταχτο κόστο του παροπλισμού του πυρηνικού εργοστασίου του Κοσλοντούι και να τη δώσει ενάψματα για την ανάπτυξη πιο φιλοπεριβαλλοντικών πηγών ενέργειας που θα περιορίζουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα πέραν του κλεισίματος ε, του πυρηνικού εργαστασίου. Αν μείνουμε λοιπόν στους στόχους της έκθεσης, ε, μπορούμε, δεν μπορούμε παρά να επενέσουμε την αρχική πρόταση και τους αξιέπαινους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα ζητήματα που έθεσε η κυρία Χάρμς είναι σημαντικά και είναι πιο γενικά και αποτελούν τη βάση για μια πολύ καρποφόρα συζήτηση για το τι ε, Πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων στην Ευρώπη, πώ θα ενισχύσουμε τη σχετική νομοθεσία. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα πυρηνική ασφάλεια. Αν όμω ε, επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα, δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε κανένα από τα ζητήματα που μα απασχολούν. Ούτε δηλαδή το συγκεκριμένο πρόβλημα του Κοσλοντούι, ούτε και την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για τις τρεις προτάσει που διατυπώνονται. Καταρχήν, το 40% των κονδυλίων χρησιμοποιείται για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η κυρία Χάρμς προτείνει να θεωρηθούν αυτά τα κονδύλια στις επενδύσεις ε, για ένα, μια νέα πυρηνική αποθήκη, αποθήκη για τα πυρηνικά απόβλητα. Και στο παρελθόν έτσι χρησιμοποιήθηκαν παρόμοια κονδύλια. Και ο πρώτος στόχος του προγράμματος ήταν να εξασφαλιστεί η συμμεταχείριση μεταξύ Σλοβακίας, Λιθουανίας και Βουλγαρίας. Και για τις δύο άλλες χώρες, Σλοβακία και Λιθουανία, έχουμε παρόμοια προγράμματα μέχρι το 2013. Οπότε, με τη χρήση των κονδυλίων αυτών ε, για τη Βουλγαρία, αντιμετωπίζεται ισότιμα με τη Σλοβακία και η Λιθουανία και η Βουλγαρία. Μετά το κλείσιμο των μονάδων 1 και 4 στο Κοσλοντούι, η Βουλγαρία θα στραφεί περισσότερο σε, ε, σε πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν περισσότερο τον άνθρακα. Τα κονδύλια της BERT στόχο έχουν τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Βέβαια, θα γίνει φέτος ε, ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το κατά πόσο αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά αυτά τα κονδύλια της ΠΕΡΤ για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι που είναι στόχος και τη Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων και της διάθεσής τους είναι επίμαχο. Δεν υπάρχει ομόφωνη γνώμη. Αλλά νομίζω θα πρέπει να συζητηθεί σε μια ευρύτερη συζήτηση. γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για να κατασκευάσουμε αυτή την αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων στην Βουλγαρία και θα χρησιμοποιηθεί και από άλλε χώρε ως προηγούμενο. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν κινητικά κονδύλια για να κατασκευάσουν αντίστοιχες αποθήκες πυρηνικών αποβλήτων. Κάτι που θα ανοίξει μια τεράστια συζήτηση. Οπότε θα δούμε τέτοιου είδους αποθήκες, πώς θα χρηματοδοτηθούν, με τι τεχνολογίες θα κατασκευαστούν. Αλλά είναι ξεχωριστό θέμα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την πρόταση για την ε, μεταφορά κτηνοβολημένων υλικών και την επαναπεξεργασία τους, νομίζω ότι το μείζον ζήτημα εδώ είναι η ασφάλεια. Και είναι πρακτικώς αδύνατο μια χώρα να καταγγείλει ή να καταστρατηγήσει τις συμφωνίες σύνδεσης. Και το νέο άνοιγμα των μονάδων 1 και 4 θα έχει τόσο αρνητικέ συνέπειε για τη Βουλγαρία που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια κυβέρνηση θα διαλέξει αυτό το νέο άνοιγμα. Σε ό,τι αφορά το, το οριστικό κλείσιμο, εδώ έχουμε και θέμα ασφάλεια και θέμα τεχνολογία, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά μέσα στη διάθεσή τη για να εφαρμόσει την, τις να υποχρεώσει την Βουλγαρία να, να τηρήσει τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συνθήκη προσχώρησης. Υπάρχει αυτό το ευρύτερο θέμα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, που είναι πολύ ευρύτερο από το Κοζιλοντούι και ίσως θα τον κόπο να το συζητήσουμε μια μέρα πιο γενικά. Ευχαριστώ κύριε Σούρουτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας που πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η κοινοτική συνδρομή για τον παροπλισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων του Κοσλαντούι. Και νομίζω ότι είναι πιστικά και τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη της χρηματοδοτικής συνδρομής της κοινότητας. Βέβαια, η έκθεση της ε, κυρίας Χάρμς τροποποιεί ριζικά σχεδόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχετικό κανονισμό. Αν γίνει διάκριση μεταξύ του πυρηνικού και του μη πυρηνικού σκέλους αυτής της ε, χρηματοδοτικής συνδρομής, διαπιστώνουμε ότι η κυρία Χάρμς Πιστεύει θα πρέπει να κλείσει το μη πυρηνικό σκέλος και να ανοίξει ένα άλλο παράθυρο της, ε, του ενταφιασμού ή της αποθήκευσης των ε, ραδιενεργών αποβλήτων ή εκτινοβολημένων υλικών. Η θέση της είναι απαράδεκτη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση αυτή. Η Βουλγαρία αποφάσισε να κλείσει τους τέσσερις αντιδραστήρες, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαβεβαίωσε ότι θα την επικουρήσει και ως προς το θέμα της, του παροπλισμού και του κλεισίματος των αντιδραστήρων, αλλά και ως προς την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών αυτού του κλεισίματος του πυρηνικού εργοστασίου. Με αυτές τις διαβεβαιώσεις έλαβε τη σχετική απόφαση η Βουλγαρία. Δεν μπορούμε να κλείνουμε εργοστάσιο παραγωγής 1.700 ΜΒ που είναι το 1 πέμπτο των, της ηλεκτροπαραγωγής της Βουλγαρίας ε, χωρίς συνέπειες ή χωρίς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις επιπτώσεις. Η κυρία Χάρμς διαπιστώνει ότι η Βουλγαρία δεν αντιμετώπισε δυσκολίες ό,τι αφορά τον εφοδιασμό της στην ηλεκτρική ενέργεια και άρα δεν αξίζει χρηματοδοτική συνδρομή για να καλύψει αυτές τις συνέπειες. Λάθος και ψεύδος, γιατί η Βουλγαρία είχε προετοιμάσει εκ των προτέρων το ενεργειακό της σύστημα για το κλείσιμο του πυρηνικού εργοστασίου του Κοσλοντούι, που είχε πολύ σημαντικές ε, δυνατότητες ηλεκτροπαραγωγής. Δεν μπορούμε να παραμελούμε και το εξή θέμα. Στην Βουλγαρία το κλείσιμο των αντιδραστήρων έγινε πολύ αρνητικά δεκτό από την βουλγαρική κοινή γνώμη. Οι σφιγμομετρήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα του βουλγαρικού πληθυσμού προτιμά το άνοιγμα του πυρηνικού εργοστασίου του Κοσλαντούι. Και ο μόνος τρόπος ε, για να δεχθεί ε, ο βουλγαρικός πληθυσμός το κλείσιμο αυτό είναι να αισθανθεί ότι υπήρξε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης. Ένα οικονομικό αντιστάθμισμα που δεν περιορίζεται μόνο στα πυρηνικά θέματα. Θέλουμε ο κόσμος να δει ποια ήταν η, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του κλεισίματος του πυρηνικού σταθμού. Και αυτό θα φανεί με έργα όπως κτίρια, υποδομές, ε, στην παιδεία, στον πολιτιστικό τομέα, στην υγεία. Θα πρέπει να φανούν αυτά τα έργα και το πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στο να αντιμετωπίσει η Βουλγαρία τη συνέπειες αυτού του κλείσιματος. Αν κλείσουμε αυτό το παράθυρο της χρηματοδοτικής συνδρομής που δεν έχει σχέση με το αμυγός πυρηνικό σκέλος του Κοσλοντούι, δεν θα καταφέρουμε να προσετεριστούμε στην ανάγκη κλεισίματος αυτού του σταθμού το βουλγαρικό κοινό που εξακολουθεί να είναι εχθρικό με αυτό το κλείσιμο. Τα 120 εκατομμύρια είναι πάνω από το 1 τρίτο της χρηματοδοτικής συνδρομής που προβλέπεται για την επόμενη περίοδο. Και η μεταφορά αυτού του κονδυλίου για την επίλυση ενός προβλήματος που θα αρχίσει να επιλύεται μετά το 2013 είναι μια δόκιμη πρόταση και δεν λύνει το πρόβλημα. ούτε συνιστά αποτελεσματική και ορθολογική χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η, πρόταση, σχετική πρόταση κυρίας Χάρμς για τη μεταφορά αυτού του κονδυλίου είναι απαράδεκτη. Στην έκθεση αναφέρεται σε πολλά σημεία η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η ανάγκη αποφυγή στήριξης ε, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν όμως παρουσιάσουμε αυτό το κονδύλιο των 120 εκατομμυρίων ευρώ ως κονδύλιο που θα αφιερωθεί στη διά, στην ε, επεξεργασία των ακτινοβολημένων υλικών θα δημιουργήσει προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι μια ενίσχυση, όχι μόνο για τη Βουλγαρία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο και ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, που έχουν κλείσει τα πυρηνικά τους εργοστάσια. Υπάρχουν και άλλες χώρες που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε να προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ισότιμα τη Βουλγαρία με τις άλλες δύο χώρες που είχαν κλείσει τα πυρηνικά τους εργοστάσια, με μια τέτοια ρύθμιση τη φέρουμε και πάλι σε άνηση θέση. Θα καταθέσουμε τροπολογίες για την έκθεση κυρίας Χάρμς και για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημένοντας τη διαφωνία μας με το περιεχόμενο της έκθεσης κυρίας Χάρμς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο ζήτημα αυτό συμφωνώ σε κάτι με την κυρία Χάμς, την κυρία εισηγήτρια. Είναι το αίτημα για την υψηλότερο δυνατό βαθμό ασφάλειας. του πυρηνικού αυτού και της διαδικασίας παροπλισμού. Τις άλλες πτυχές διαφωνώ πλήρως. Γιατί όπως έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία ένταξης ε, της Βουλγαρίας δεν συμπεριελάμβανε μόνο το κόστος ε, του παροπλισμού αλλά και αποζημίωση για την απώλεια παραγωγικής δυνατότητας. Και δεν ήταν μόνο το θέμα η ενεργειακή ασφάλεια της Βουλγαρίας, αλλά και γειτονικών χωρών, γιατί η Βουλγαρία εξήγαγε και σε άλλες ε, χώρες, όπως τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Πούγουδουμού. Και και βεβαίως μετράει και για τον ε, προϋπολογισμό μας, το έχουμε υπολογίσει και είναι προφανές πως είναι ευάλωτη αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία κοινωνικά και δεν μπορούμε να ε, διακινδυνεύσουμε τις χώρες ε, τις γειτονικές μας στα Βαλκάνια. Χρειαζόμαστε σταθερά Βαλκάνια και δεν πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές στην Ευρώπη. Γιατί χωρίς τα Βαλκάνια δεν είναι πλήρης η Ευρώπη πρέπει να υπάρχουν ή να υπάρχει ήπια και ήρεμη εμπλοκή των Βαλκανίων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω εδώ πέρα η Βουλγαρία θα αποτελέσει το βασικό δείγμα. Προετοίμασα λοιπόν 8 τροπολογίες στο κείμενο και ηρεμη μπλοκή των βαλκανιων στην ευρωπαικη ενωση και νομιζω εδω περα η βουλγαρια θα αποτελεσει το βασικο δειγμα προετοιμασα λοιπον 8 τροπολογιες στο κειμενο και ελπιζω πως ε, η προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει δεκτή από το Κοινοβούλιο. Και ελπίζω να γίνει ε, δεκτή και η αποζημίωση. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. έχουμε οδυνηρές ε, αναμνήσεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση. Και επομένως ρωτώ το εξή. Ε, είμαστε βέβαιοι ότι εμείς σαν κοινοβούλιο έχουμε δυνατότητα ελέγχου ε, των κονδυλίων αυτών. Και δεύτερη ερώτηση, η οποία απευθύνεται στην ε, Επιτροπή. Έχουμε διασφάλιση ότι για την χρήση των κονδυλίων αυτών ε, και όσον αφορά την εξέβρεση των καταλλήλων εταιριών θα υπάρχει διαφάνεια. Τρίτον, ε, θα ε, υπάρξει η έννοια κοινοτικής προτίμησης όσον αφορά αυτήν την αποδέσμευση του χώρου. Bedanke mich sehr. Darf ich der Kommission Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στην Κομισιόν, κ. Φάρος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισηγήτρια για την ε, έκθεση αυτή. Βλέπω μεγάλη ικανοποίηση πως ε, υπάρχει αρκετά μεγάλη σύγκληση μεταξύ της υποβληθής σας έκθεσης ε, και της πρότασης της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα και ε, στα δύο έγγραφα αναγνωρίζεται πως πρέπει να συνεχιστεί ο παροπλισμός και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές και στις δύο έκθεσεις αναγνωρίζεται πως μέχρι το 2013 πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και πως η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του σχετικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Επίσης έχουμε συμφωνία για την τάξη μεγέθους ε, της χρηματοδότησης ε, που απαιτείται γιατί και η συγγήτρια θεωρεί πως 300 ε, εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια είναι ε, το σωστό ποσό ο συνολικό πακέτο. Κατόπιν έχουμε το κρίσιμο σημείο που υπάρχει κάποια απόκληση και αυτό είναι το θέμα πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Θεωρώ πως ε, για τα 180 εκατομμύρια του παροπλισμού συμφωνεί και η συγκήτρια. Οπότε το ζήτημα είναι τα 120 εκατομμύρια, το εάν προβλέπετε να χρησιμοποιηθούν όπως είναι στο άρθρο 30 της Συνθήκης Ένταξης για έργα ενέργειας ή εάν θα πάνε τα 120 εκατομμύρια για ένα σχέδιο τελικής αποθήκευσης στην Βουλγαρία για τα εξαντλημένα καύσιμα. Πρώτα απ' όλα να διαβεβαιώσω την εισηγήτρια πως ε, η Κομισιόν ε, θεωρεί πως ε, οι τελικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις έχουν εξίσου μεγάλη πολιτική σημασία για εμάς και πως ο κύριος Έτιγκερ, ο Επίτροπος, είπε πως η Κομισιόν για το ζήτημα αυτό η κυρία Έτιγκερ με συγχωρείτε, είπε πως σκοπεύει να υποβάλει μια τέτοια πρόταση. Βεβαίως το ζήτημα τίθεται εάν είναι σωστό, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο στην πρόταση, να προδικάσουμε από τώρα την χρηματοδότηση τέτοιων έργων με βάση μία πρόταση παροπλισμού που δεν έχει σχέση με την τελική διάθεση των αποβλήτων η Επιτροπή νομίζω πρέπει να θέσει το ερώτημα το εάν με μια τέτοια συμπεριφορά προκαλέσουμε μια βάδα και ανοίξουμε την πόρτα έτσι ώστε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που θίγονται από τον παροπλισμό ζητήσουν και αυτά κοινοτική χρηματοδότηση. Αυτό όμως δεν απαντά το ερώτημα της προσέγγισης, δηλαδή εάν έχουν νόημα τα έργα ενέργειας. Και εδώ πέρα θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Τα ενεργειακά έργα στην Βουλγαρία δεν σημαίνουν μόνο νέες δυνατότητες παραγωγής. Με το κλείσιμο του Κοσλοντούι, έχουμε αλλάξει δραστικά την δομή της παραγωγής. Γνωρίζουμε λοιπόν πως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις για να καλυφθεί το νέο τοπίο, η νέα κατάσταση. Γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη πως κάποιοι σταθμοί μετασχηματισμού πρέπει να αποκτήσουν περαιτέρω επενδύσεις για να έχουμε μια σταθερή ροή ηλεκτρισμού τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν ούτω ή άλλω, ανεξαρτήτως του εάν χρειάζονται περαιτέρω δυνατότητε παραγωγή ή όχι. Και όσον αφορά δε τα έργα ενεργειακή αποτελεσματικότητας, εκεί πέρα υπάρχει διχογνωμία. Κατά την απόψή μας και σύμφωνα με την αξιολόγησή μας, η Βουλγαρία είναι ένα κράτος μέλος το οποίο χρησιμοποιεί, ε, έχει 8 φορές μεγαλύτερη ένταση ενέργειας από τον κοινοτικό μέσο όρο και εδώ πέρα μπορούν ακριβώς να γίνουν οι μεγαλύτερες οικονομίες. Και εδώ πέρα έχει νόημα να γίνουν οι επενδύσεις. Εγώ ευχαριστώ ε, να σας δείξω μία έκθεση ανεξαρτήτων συμβούλων για το πώς αξιολογούνται αυτές οι επενδύσεις και σε ποια εξαιρετικά αποτελέσματα καταλήγουν. Το θέμα της διάθεσης των κονδυλίων είναι πράγματι αιτιολογημένο, γι' αυτό εμείς προτείναμε να πάνε μέσω ενός ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η ροή αυτή θα ελέγχεται τακτικά, τα έργα θα υποβάλλονται σε μια επιτροπή που θα τα εξετάζει λεπτομερώς. Διαφάνεια, έλεγχος είναι δεδομένα και μπορώ να σας υποσχεθώ πως αυτή τη στιγμή το ελεγκτικό συνέδριο αυτή τη στιγμή ε, ε, κάνει έναν έλεγχο της απόδοσης. Συμπέρασμα. Τι ζητάει η Κομισιόν. Μην προδικάσουμε πού θα πάνε τα λεφτά, εάν θα πάνε σε τελική αποθήκευση και να επενδύσουμε σε ενεργειακά έργα που έχουν νόημα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν στον τομέα του δικτύου και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ähm, σας ευχαριστώ. Νομίζω θα δεχτούμε την ε, προσφορά σας και θα ήθελα να μας δώσετε αυτή την ε, έκθεση πράγματι. κυρία Χάρμς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον του να ξοδευτούν περισσότερα λεφτά στη Βουλγαρία για ενεργειακή αποδοτικότητα και για μια υφόρο στρατηγική. Απλά διαπιστώνω πως ε, με βάση τα όσα γνωρίζω η σχέση μεταξύ των εξόδων που κάνει από ίδια μέσα η Βουλγαρία στον τομέα αυτών και της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το Ταμείο Αυτό Παροπλισμού μάλλον ε, μας λέει πως ε, η Βουλγαρία δεν έχει κάνει κεντρική ενεργειακή πολιτική την ενεργειακή αποτελεσματικότητα οπότε όσο καλά και αν είναι τα μεμονωμένα έργα που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να το λάβει υπόψη ε, στη συνολική αξιολογική της η Κομισιόν γιατί ακόμα είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε αυτό το άλμα αποτελεσματικότητας στην ε, Βουλγαρία. Έτσι εκτιμώ εγώ τη σημερινή κατάσταση και τα πράγματα μπορούν μόνο να βελτιωθούν. Δεύτερον, τα Βεβαίως ως πράσινοι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να ενισχύσω είτε τις ρωσικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία είτε γενικά την ατομική ενέργεια και να τους δώσουμε λεφτά για να διαθέσουν τα απόβλητα. Από την άλλη όμως τα πράγματα έχουν ως εξής. Αν εμείς ως Ευρωπαίοι δεν σταθούμε όχι μόνο στα οικονομικά αλλά και στις προδιαγραφές ασφαλείας και δεν αναλάβουμε την ευθύνη για την ασφάλεια στον παροπλισμό του Κοσλοντούι πρέπει να δούμε και την συνολική κατάσταση. Και δεν ξέρω τι έχει συμπεράνει η Κομισιόν από τη Βουλγαρία, αλλά εγώ δεν έχω την εντύπωση πως ε, η Βουλγαρία έχει, έχει προετοιμαστεί όσον αφορά τη στρατηγική παροπλισμού και διάθεσης των αποβλήτων και η αιτιολόγηση είναι οι συμβάσεις ε, με την Ρωσία που μας τις έδωσε η Κομισιόν. Είναι στην έκθεση για την κοινή σύμβαση λέει πως δεν υπάρχουν επαρκή μέσα για την τελική αποθήκευση στη Βουλγαρία και πως η επανεπεξεργασία στη Ρωσία είναι ένας ε, τρόπος ο οποίος ε, θα επιβαρύνει υπερβολικά τις μελλοντικέ γενναίες. Δεν συμφωνώ εγώ γιατί η επανεπεξεργασία ειδικά στη Ρωσία, τόσο πάμε πάρα πολύ μακριά στη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω πως ε, αποφεύγουμε έτσι την επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών. Σημαντικό για μένα είναι πως οι ίδιοι οι Βούλγαροι λένε πως δεν έχουν λεφτά για να προετοιμάσουν την τελική αποθήκευση, γι' αυτό εξάγουν το ε, χρησιμοποιημένο κάψιμο ε, προς τη Ρωσία. Είναι μια κατάσταση την οποία εγώ δεν αποδέχομαι και κατά την άποψή μου, ειδικά αν ο κύριος ε, Έτιγκερ ε, ε, θεωρεί πως θα πρέπει να τα εξαγάγουμε αυτά για να τα αποθηκεύσουμε φτηνά, δεν το θεωρώ αποδεκτό. Και αυτό το κάνει η Βουλγαρία και θα το κάνουν και άλλες χώρες. Δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Η προσφορά για αυτά τα 120 εκατομμύρια να πάνε σε ένα ταμείο το οποίο πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο βεβαίως αν είναι να μιλήσουμε για ασφαλή διάθεση ε, νομίζω πως θα πρέπει να την ζυγίσουμε αυτή την επιλογή για να δούμε ε, να τη ζυγίσουμε έναντι του ποια άλματα μπορούν να γίνουν στα αποτελεσματική χρήση ενέργειας αλλά θα δούμε βεβαίως και την συζήτηση με βάση τροπολογία που θα κατατεθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, έντονη αυτή συζήτηση. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο. Τροπολογίες μέχρι τις 4 Μαρτίου. 18 δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. 19 γνωρίζετε, έχετε τις επόμενες ημερομηνίες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο λοιπόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη σημερινή συζήτηση και σας εύχομαι μια ενδιαφέρουσα ημέρα. Γεια σας.